miserable day. I'm sure you understand. <laughs> so, let's go. Thank you. Thank you for being... Ας ξεκινήσουμε και σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Όλοι σας. Ευχαριστούμε. Και τον κύριο Πίστερ Χάστινγκς από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ε, εποπτείας προσωπικών δεδομένων που είναι εδώ κοντά μας. Για το σημείο 14 με την αναδιατύπωση της εκθέσεως, με την έκθεση πάνω για την αναδιατύπωση τη πρόταση για τη δημιουργία του συστήματο Eurodac για τη σύγκριση φιλικών αποτυπωμάτων με την κυρία Μακοβέη, η οποία δυστυχώ δεν μπορεί να έρθει σήμερα εδώ. Θα την αντικαταστήσει ο κύριος Δοφός. Κύριος Πέτερ Χάστινγκς. Θα μιλήσει, μετά θα μας ενημερώσει η Κυπριακή Προεδρία. Και θα ανοίξει η συζήτηση. Ξεκινάει όμως ο κύριος Φως πρώτος, εκπρόσωπος της εισηγητρίας. Πρόεδρε, θα σας παρουσιάσω εγώ την ε, έκθεση της ε, κυρίας Μακοβέη, η οποία καλωσορίζει την υποβολή των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κανονισμός Eurotac είναι... Α, είναι ένα πολύ σημαντικό πακέτο και έχει φυσικά πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει για την αντιμετώπιση των πολλαπλών ε, προτάσεων για χορήγηση ασύλου. Έχουμε λοιπόν την δυνατότητα οι αρχές επιβολής της τάξης ε, στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορούν να επιβάλλουν σύγκριση τακτηλικών αποτυπωμάτων που που διακρατούνται στη Γιούροντα, καλά μόνο ότι υπάρχει υποψία για πολύ σοβαρά εγκλήματα και οργανωμένη εγκληματικότητα και σε πολυορισμένη βάση. Η συμφωνία αυτή αποτέλεσε μια ισορροπημένη ε, λύση που προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις για το Ευρωπαϊκό Πακέτο Ασύλου με την ε, συνολική πρόταση του 2012 όπως άλλωστε εξηγεί Mm-hmm. Όπως άλλωστε εξηγεί στο, στο, στο επεξηγηματικό μνημόνιο η Επιτροπή. Κυρία Μακοβέ, λοιπόν, καταθέτει μια σειρά από τροπολογίε, όπως προτείνεται. Τεχνικού χαρακτήρα τροπολογίε, προτάσει για την πρόταση αναδιατύπωση. εσωτερικές αναφορές, με στόχο την διευκρίνηση του κειμένου, παραδείγματι, αντικατάσταση του όρου technology από τον όρο technics στο σημείο 4 και στο άρθρο 4 τον, ε, την αναφορά σε μια μεταβατική περίοδο και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη διάρκεια αυτής και το δικαίωμα της πρόσβασης στα δεδομένα. Άλλες τροπολογίες στόχο έχουν να συμπεριλάβουν προτάσεις, ε, εύστοχες προτάσεις Ευρωπαϊκής Αρχής Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων με στόχο τη βελτίωση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων επί παραδείγματι. Η πρόσβαση στην η, πρό... η πρόσβαση των διοκτικών αρχών ε, υπόκειται. Ναι, δεν ξέρω αν μπορώ να προφέρω αυτές τις λέξεις, λέει ο κύριος Φως. Ε, υπόκειται λοιπόν σε αυστηρές προδιαγραφέ και στην ε, ε, διερεύνηση μέσα από μια βάση δεδομένων με αρνητικά αποτελέσματα, την εξαντλητική εξέταση ενός ερωτηματολογίου και με την προϋπόθεση επίσης κινδύνου τρομοκρατικών δραστηριοτήτων, προετοιμασίας τους, οργάνωσής τους, υλοποίησής τους, εφόσον βεβαίως υπάρχει δυνατότητα συγκρισιμότητας χρήσιμη με τη βάση δεδομένων της Eurodac. Χρήσιμες με την έννοια ότι μπορεί να αποτραπούν, να προληφθούν ε, κάποιες από τις εγκληματικές δραστηριότητες και δεύτερον απαιτούνται τα εξής ε, βήματα για την πρόσβαση. Πρώτον, υποβολή ε, ηλεκτρονικού αιτήματο από τι αρμόδιε αρχέ. Δεύτερον, επαλήθευση του αιτήματο από τι επαληθεύουσε αρχέ. Τρίτον, οι επαληθεύουσε αρχέ θα πρέπει να διαβιβάσουν το αίτημα στην εθνική, στο Εθνικό Σημείο Πρόσβαση. Και σε περίπτωση επιτυχούς εντοπισμού δεν αποκαλύπτεται το πρόσωπο του εμπλεκομένου προσώπου στις αρχές Σημειώνει δε η εισηγήτρια ότι είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο να τηρήσει προηγούμενη ε, δέσμευση για την ε, δέσμη μέτρων σχετική με το άσυλο και να προχωρήσει ταχύτατα στην έκθεση αυτή, έτσι ώστε να γίνει μια πρώτη ψηφοφορία προς ανατολισμού στην Επιτροπή μας στη συνεδρίαση της 17ης-18ης Οκτωβρίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα, ας ακούσουμε τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εάν έχει κάποια σχόλια αφού άκουσε την παρουσίαση της εκθέσεως. Παρακαλώ. Thank you very much, Mr. Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είμαι θα ευγνώμονες για την ε, εργασία της εισηγητρίας. Η Κομισιόν μπορεί να δεχτεί κάποιες πρακτικής φύσεως τροπολογίες. Είχαμε και μια αντίστοιχη ε, συζήτηση με το Συμβούλιο άλλωστε και πρέπει να δούμε και ποιες ε, είναι οι περαιτέρω τροπολογίες οι οποίες ε, ενδεχομένως μπορούν να ενσωματωθούν στον επερχόμενο τριμερή διάλογο. Γνωρίζετε ότι πρόθεση όλων είναι να υπάρχει έγκριση για το κοινό σύστημα ασύλου μέχρι το τέλος του, ε, συστήματος, ε, το τέλος έτους και ελπίζουμε ότι και το Κοινοβούλιο θα συμβάλλει έτσι ώστε ε, να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τα ζητήματα αυτά όσο γίνεται πιο γρήγορα και βεβαίως προσδοκούμε να έχουμε και μελλοντική καλή συνεργασία και με την εισηγήτρια και τους σκιώδες. Ευχαριστώ πολύ. Η Κυπριακή Προεδρία παρακαλώ η Κυπριακή Προεδρία. Παρακαλώ. Thank you, Chair. Thank you for the honor. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε να τους καλείτε. Όπως μάλλον γνωρίζετε, η Επίτροπη Μονίμων Αντιπροσώπων συζήτησε και υιοθέτησε με επαρκή πλειοψηφία την εντολή για το Συμβούλιο. Θεωρούμε ότι το κείμενο που υιοθετήθηκε εχθές συμπεριλαμβάνει συνεπάγεται σημαντική προσθέμενη αξία μετά τις συζητήσεις των εργασίας του Συμβουλίου και μπορεί να αποτελέσει μια βάση για ε, κίνηση άτυπου διαλόγου με το Κοινοβούλιο. Και ευχαριστώ την εισηγήτρια για την έκθεσή της, θα θέλω να επισημάνω ότι η Eurodac είναι το τελευταίο κομμάτι που λείπει από το Ευρωπαϊκό Κοινό Σύστημα Ασύλου, που ελπίζουμε τουλάχιστον σιγά σιγά παίρνει σάρκα και οστά. Η Eurodac νέο κείμενο μεν, αλλά το τέταρτο στη σειρά κείμενο μετά το 2008 αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό τη δουλειά που έχει μέσω μεσολαβήσει από το Δεκέμβριο του 2008 με την πρώτη πρόταση και όπως είπαμε όπως υπόθηκε, εξασφαλίζει μια περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης για τις διοκτικές αρχές στην περίπτωση προσπαθειών πολέμηση οργανωμένου εγκλήματος τρομοκρατίας. Ως Προεδρία, ιδιαίτερως είμαστε ικανοποιημένοι για το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την πρόθεση να τηρήσει το στόχο της ολοκλήρωσης του πακέτου για το άσυλο μέχρι τα τέλη του έτους. Έχουμε εργαστεί ουσιαστικά σε άλλα Έχουμε συνεργαστεί ουσιαστικά σε άλλα ε, στάδια αυτής της προσπάθειας για το Δουβλίνο και για άλλα και δεδομένη και τη αποφασιστικότητα του Συμβουλίου, πιστεύουμε ότι θα μπορούσαν να ξεκινήσουν το χειρότερο δυνατό οι τριμερεί διαπραγματεύσει, έτσι ώστε να ε, τηρήσουμε τον στόχο αυτών μέχρι το τέλο του έτου δηλαδή τη έγκριση. Τόσο η Προεδρία όσο και τα κράτη-μέλη καταβαλούν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τιμήσουν την κοινή αυτή πολιτική δέσμευση και επαναλαμβάνω για μια φορά ότι είμαστε ευγνώμονες για τη μέχρι τώρα συνεργασία. Και θα θέλαμε να τη συνεχίσουμε με, την ίδια, ε, με τον ίδιους ρυθμούς μέχρι και το τέλος του έτους. Ε, ευχαριστώ και τώρα ο κύριος Χάστινγκς, ο οποίος έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου προσφέρετε να σας παρουσιάσω τη γνωμοδότηση που σας έχουμε αποστείλει στις αρχές Σεπτεμβρίου. Δεν είναι η πρώτη γνωμοδότηση. Κάποιοι την έχουν αναφέρει ως ιστορικό στοιχείο. Δύο γνωμοδοτήσεις, μία του 2000, μέσα του 2009, μια θετική αποτίμηση καταρχάς ε, για, την, ε, για τον κανονισμό Eurodac και άλλη η μία έκθεση, μάλλον επικριτική ως προς το δικαίωμα πρόσβασης, το 2009 όλα αυτά. Εκ τότε όμως πολλά σημαντικά πράγματα έχουν δεσολαβήσει, εκ των οποίων ορισμένα, ε, όπως η θέση λειτουργία της συνθήκης της ε, Λισαβόνας, της συνθήκης Λισαβόνας έχουν αλλάξει ουσιαστικά τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα των θεμελιωδών ε, ελευθεριών και ακούσαμε τον ε, Επίτροπο, την Επίτροπο των Αρμόδια για Ανθρώπινα Δικαιώματα να μιλάει για μηδενική ανοχή σε παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου λοιπόν πρέπει να πω ότι με κατάπληξη διαπιστώνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να μην τηρήσει την πολιτική της στην περίπτωση αυτή, δηλαδή την ε, πολύ ε, επικριτική αξιολόγηση συνεπειών ε, της πολιτικής αυτής που γίνεται στο παρελθόν. Δεν θα γίνεται, δεν, θα, δεν μπορούν να κρυθούν ικανοποιητικέ οι προηγούμενες αξιολογήσεις για λόγους που έχω ήδη εξηγήσει και έτσι θα ήθελα να επισημάνω ότι δυστυχώς η Επιτροπή σας δεν είναι σε θέση να προβεί σε πλήρη αξιολόγηση αυτού του κρίσιμης σημασίας, κέρια σημασίας ε, νομοθετήματος για το, τα πιο κρίσιμα θέματα πρόσβασης ε, της ε, δίωξη στα προσωπικά δεδομένα και θα ήθελα να υπογραμμίσω, όπως άλλως το πράξαμε και στην ομοδότηση, ότι αντιλαμβάνομαι βεβαίω πως το να υπάρχει μια βάση δεδομένων με δακτυλικά αποτυπώματα μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη ως συμπληρωματικό μέσον σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά δεν εξετάζεται αν πρέπει να είναι χρήσιμο γιατί εγώ εδώ έχουμε να κάνουμε χωρίς ουδεμία αμφιβολία με παραβίαση της, ε, των δικαιωμάτων των εμπλεκομένων ανθρώπων και με τους περιορισμούς που έχει επιβάλει ο νόμος. Θα πρέπει να εξετάσουμε αν είναι απαραίτητη και αναλογική η χρήση αυτού του μέσου. Ε, από αυτό αποδιαπιστώνουμε λοιπόν όχι μόνο δεν αρκούν, αλλά του εναντίον τίποτε δεν επαρκεί ώστε να δείξει ότι είναι αναλογική η αξιοποίηση, δεν υπάρχει ανάλυση, δεν προσφέρονται εναλλακτικέ επιλογές, όπως υφιστάμενα μέσα νόμιμα, επί παραδείγματι άλλη πρόσβαση σε δακτυλικά αποτυπώματα. Και θα έλεγα ότι η αναγκαιότητα δεν είναι το να συμπληρώσουμε ακόμη ένα κομμάτι στο πλέγμα ε, σχέσεων με το Συμβούλιο, στο πλέγμα νομοθετημάτων. Αυτή η ιδέα μπορεί να οδηγήσει σε λάθος συμπεράσματα. Και ξέρω ότι είναι πολύ σκληρή η γλώσσα που χρησιμοποιώ. Εδώ λοιπόν τώρα αυτό που συμβαίνει είναι ότι θα έχουμε ένα εργαλείο που μπορεί να υιοθετηθεί και που θα στοχεύει μόνο όποιον έχει καταθέσει αίτημα για άσυλο, για χορήγηση ασύλου. Αν δηλαδή σε μία σκηνή εγκλήματος ε, καταγραφεί δακτυλικό αποτύπωμα, μπορεί ένα ετών το άσυλο να εντοπιστεί μέσω αυτή τη βάση τη και ενώ όλοι οι λοιποί εμπλεκόμενοι δεν θα μπορούν να εντοπιστούν γιατί δεν θα έχουν ε, εκτεθεί τα αποτυπώματά του στον έλεγχο των, στην επαλήθευση από τι αρχέ. Η πίεση λοιπόν, οι ε, προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Συμβουλίου για να προωθηθεί αυτό το μέτρο αποτελεί ένα κλασικό παράδειγμα χρήση δεδομένων που τυχαίω υφίστανται για άλλο λόγο, για άλλο σκοπό. Γιατί η βάση αυτή συστήθηκε με πολύ αυστηρού ε, όρου και προδιαγραφέ, ε, να μην χρησιμοποιούνται τα δεδομένα αυτά παρά μόνο για λόγου ασύλου και αυτέ οι προποθέσει θα πρέπει να τηρηθούν. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει. Εάν λοιπόν ο νομοθέτης τυχόν αποφασίσει για λόγους που ανήκουν στη διακριτική του ευχαίρεια να ρυθμίσει κατά τρόπο θεμητό το νομοθέτημα αυτό, χρειάζονται, πιστεύω, περισσότερες διαφορετικές διασφαλιστικές δικλείδες. Επί παραδείγματι. Επί παραδείγματι, δεν μπορεί να βοηθήσει στην προαγωγή των ε, ερευνών. Εάν κανεί, σε παραδείγμα, έχει ένα κατάλογο από τον οποίο μπορεί να διαγράψει κάποιου υποτιθέμενου υπόπτου, ε, θα μπορούσε βεβαίω να προχωρήσει τι ερευνέ του. Αλλά το κείμενο δείχνει ξεκάθαρα την υποψία που εκφράζεται ότι ο ε, φυσικός αυτούργος μιας τρομοκρατικής επίθεσης ή μιας ε, σοβαρής εγκληματικής ενέργειας, ο δράστης, έχει ήδη υποβάλει έτοιμα για άσυλο. Με αυτή την προϋπόθεση ξεκινάει. Μα η επαλήθευση πρέπει έπρεπε να γίνεται πραγματικά ανεξάρτητα από ανεξάρτητη αρχή, από δικαστική αρχή συγκεκριμένα, κατά προτίμηση. Και έτσι λοιπόν, εάν ε, διατρέξουμε τους όρους και βέβαια Αναγνωρίζω ότι με πολύ μεγάλη προσοχή έχουν καταγραφεί οι αυτοί, αλλά αν τους διατρέξουμε καταλήγουμε στο συμπεράσμα ότι δεν αντέχουν στην επαλήθευση της, ε, ε, των διασφαλιστικών δικλείδων, δηλαδή της αναλογικότητας και όχι υπερβολικής παραβίασης των δικαιωμάτων. Εδώ λοιπόν, όπως είπα και την προηγούμενη φορά, έχουμε να κάνουμε με μία υφέρπουσα διάβρωση των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Και έτσι. Προτείνω. Η συγγετρία όχι μόνο να λάβει υπόψη, όπως αναφέρθηκε στα τέλη της εκθέσεως, κάποιες εύστοχες παρατηρήσεις, αλλά να καλύψει το πιο σημαντικό ζήτημα που προκύπτει και να δώσει, να δώσει η Επιτροπή σας, μια πιστική απάντηση, είτε επί το θέμα των αρχών, είτε επί το θέμα των δικλείδων των διασφαλιστικών. Και κλείνοντας, υπάρχει μια σειρά πρόσθετων προτάσεων σε βαθμό λεπτομέρειας, για τις οποίες εάν δοθεί περισσότερο περιθώριο μελέτης και, ε, και με κάποιες τροπολογίες θα μπορούσαν ενδεχομένω να γίνουν δεκτές. Αλλά εγώ στον χρόνο που έχω στη θέση μου τώρα θέλω να επικεντρωθώ μόνο στο σοβαρό ζήτημα που έχουμε ενώπιόν μας και τελικά ε, συνοψίζεται στο εάν χρειάζεται, εάν αναλογικά είναι απαραίτητο να ε, γίνει η χρήση αυτών των δεδομένων. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να επαληθευθεί αν, υπάρχει η προδιαγραφή, αν τηρείται η προδιαγραφή τη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εάν είναι αναγκαία και αναλογική ή ε, αναγκαίο και αναλογικό ο παραμερισμό των δυσφυλιστικών δικλείδων που έχουμε εδώ και 10 περίπου χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χάστινγκ. Θα έχουμε τώρα μια πρώτη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 στον γύρο των διαπραγματεύσεων Eurodac. Και όταν έπρεπε να εξηγήσουμε στους υπολείπους ε, γιατί έπρεπε να ε, δώσουμε την άδεια να ληφθούν ε, τα δακτυλικά αποτυπώματα από τους ετούντες άσυλο. Κάναμε πολύ προσπάθεια να το εξηγήσουμε. Εγώ στήριξα την πρόταση αυτή γιατί ε, όταν, υπάρχει, όταν υπάρχουν διπλή κατάλογοι χρειάζεται και κάποιος έλεγχος. Αλλά δεν ήταν κάτι που θα γινόταν αυτόματα. Εάν ξέραμε στις πρώτες διαπραγματεύσεις ότι αυτό το σύστημα ε, θα χρησιμοποιείται για την επιβολή του νόμου, δεν νομίζω ότι θα είχε συζητηθεί ποτέ αυτό το ενδεχόμενο, γιατί ήταν απολύτως αντίθετο προς το πνεύμα των διαπραγματεύσεων. Επομένως, πρέπει κανείς να έχει εξαιρετικά καλή επιχειρηματολογία, έτσι ώστε να αλλάξει την φύση ενός ήδη πολύ ευαίσθητου εργαλείου. Και στην ομάδα μου και πάντα προσπαθώ να είμαι πρακτική θετικό πνεύμα, ε, να ε, δείχνω κατανόηση και προς τα θέματα της επιβολής του νόμου και ε, του εγκλήματος, του ιδιαίτερου επαχθών εγκλημάτων κτλ. Αλλά παρόλα αυτά εδώ πάμε πάρα πολύ μακριά. Συμφωνώ απολύτως με κάθε λέξη που είπε ο κύριος Χέντριξ. Νομίζω ότι θα πρέπει, συγγνώμη, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ε, προσεκτικοί. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ζητήσουμε την Επιτροπή ε, να ε, μας δώσει σωστή επιχειρηματολογία. Εντάξει, το Συμβούλιο το θέλει, αλλά θα πρέπει να μας πει κιόλας ε, πόσες είναι οι υποθέσεις οι οποίες δελευκάνθηκαν ε, λόγω της ε, χρήσης αυτών των αποτυπωμάτων. Και δεν νομίζω ότι υπάρχουν πιστικά επιχειρήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Έστω και αν υπήρχαν αποδεκτικά στοιχεία, θα ήταν πολύ δύσκολο παρόλα αυτά να βρεθεί μια έτσι ισορροπημένη θέση, γιατί ε, θα ε, μπορούσε εύκολα να στιγματιστεί κατά κάποιο τρόπο αυτό το σύστημα ε, το οποίο δημιουργείται για τους ετούντες άσυλο και που μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή για επιβολή νόμου. Δηλαδή γιατί μονάχα οι ετούντες άσυλο να έχουν ένα τέτοιο μητρό αποτυπωμάτων και να μην πρέπει όλοι οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης να δώσουν τα αποτυπώματά τους έτσι ώστε δυνητικά να χρησιμοποιηθούν για την επιβολή του νόμου. Είμαι μάλλον πεπισμένος ότι η κυρία Μακοβέη έχει κάνει πάρα πολλά καλά πράγματα στο Κοινοβούλιο, αλλά δυστυχώς αυτή τη φορά ενδεχομένως η ομάδα μου θα ζητήσει απόρριψη χωρίς κανένα ελαφρυντικό. Και στρέφομαι και προς το Συμβούλιο για να του πω το ίδιο πράγμα. Δεν είναι δυνατόν να δούμε μονάχα αυτό το ζήτημα και να αφήσουμε όλα τα άλλα τα οποία συνδέονται με το άσυλο. Ε, θα πρέπει να υπάρχει μία δέσμη. Και ακόμα και αν υπάρχει δέσμη, φοβούμε ότι παρόλα αυτά δεν θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, η κυρία Κέλλερ. Thank you very much. Um, thank you. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χάστινγκ, για τη ε, διαφωτιστική σας παρουσίαση. Είπατε, ε, θέσατε κάποια ερωτήματα τα οποία και εμείς θέλουμε να θέσουμε. Βλέπω αυτό το σύστημα Eurodac και αναρωτιέμαι γιατί θέλουν αυτή την πρόσβαση οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Δηλαδή γιατί ε, δυνητικά θα υπάρχουν περισσότεροι ας πούμε τρομοκράτες ε, στο, μεταξύ των ετούντων άσυλο και όχι ε, στον υπόλοιπο πληθυσμό. Θα πρέπει να είμαστε σαφείς εδώ. Επίσης και όταν ζητήσαμε και από τη Europol να μας δώσει κάποια στοιχεία επί των οποίων βασίζονται για το αίτημά τους αυτό δεν ήταν σε θέση να μας δώσει. Θα μπορούσατε λοιπόν να μου ξεκαθαρίσετε αυτό το ζήτημα, γιατί πρέπει να έχουμε στοιχεία, πρέπει να έχουμε ε, ε, ε, πιστική επιχειρηματολογία, θέλουμε αποδεικτικά στοιχεία, θέλουμε αποδείξεις. Δεν είναι δυνατόν να ε, ε, παραβιάζονται θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα χωρίς λόγο και αιτία. Επίσης δεν νομίζω ότι μεταξύ των ε, ετούντων άσυλο κινδυνεύουμε να βρούμε περισσότερους τρομοκράτες από ό,τι στον υπόλοιπο πληθυσμό. Οι ετούντες άσυλο πάντως θα είναι η μόνη ομάδα η οποία δίνει τα δακτυλικά της αποτυπώματα και τα δακτυλικά της αποτυπώματα θα πρέπει να ε, εξετάζονται για το κατά πόσον συνδέονται με τρομοκρατικές ενέργειες ή όχι. Ε, δηλαδή τους αντιμετωπίζουν, τους σε άσυλο σαν ε, δυνάμοι εγκληματίες Κάθε φορά δηλαδή που έχουμε ένα πρόβλημα, μια εγκληματική ενέργεια, τρομοκρατική κτλ. Ε, θα γίνεται προσπάθεια, θα λένε ε, πάντα ας ελέγξουμε και τον κατάλογο των ετούντων άσυλο. Ε, είναι σαν να τους εγκληματοποιούμε εξ αρχής. Και επίσης δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε νομοθεσία για την οποία και νομοθετήματα για τα οποία δεν έχει υπάρξει καμία μελέτη αντικτύπου και που ε, ταυτοχρόνως παραβιάζουν παράφορα συγγνώμη, κατάφορα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης όλοι μιλούν για συμφωνία, για deal, αλλά η δέσμη του ασύλου έχει ξεκινήσει πριν από καιρό και έχει αποτύχει για την ώρα και δεν είναι φταίει γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίσαμε ήδη το 2009 για το άσυλο ε, και ε, για ε, τέσσερα χρόνια μπλοκάρισε το Συμβούλιο το θέμα αυτό. Δεν είναι δικό μας λοιπόν. Τώρα μας λένε δεν, δεν υπάρχει χρόνος. Ναι, αλλά δεν φταίμε εμείς γι' αυτό. Και η, η πρόσβαση της αστυνομίας θα σήμαινε άρση ε, ε, της ε, ρήτρας αλληλεγγύης του Δουβλίνου. Δεν υπάρχει όμως τέτοιος εναιρετικός μηχανισμός στο, στη Συμφωνία του Δουβλίνου. Και εν πάση περιπτώσει όλη η νομοθεσία για το άσυλο αφορά το άσυλο και αφορά τους ετούντες άσυλο. Δεν αφορά ούτε το έγκλημα ούτε την τρομοκρατία. Τέλος, θα συμφωνήσω απολύτως με αυτά που είπε ο κύριος Χάστινγκς όσον αφορά τον περιορισμό του πεδίου. Εμείς είμαστε πάντα πάρα πολύ προσεκτικοί και ε, διαρκώς όμως ζητούμε όλο και περισσότερα στοιχεία. Ε, τώρα υπάρχει δυνατότητα ε, να παίρνει κανείς στοιχεία και δακτυλικά αποτυπώματα και από τρίτες χώρες. Αλλά αυτή η, ε, αυτή η πολιτική δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Και από τη στιγμή που δεν έχουν γίνει μελέτε επιπτώσεων, από τη στιγμή που δεν μπορείτε να μας υποβάλλετε και να μας παρουσιάσετε κάποια αποδεκτικά στοιχεία, δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε μια τέτοια κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Η, κυρία Λάτφορντ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνώ με τα σχόλια των συναδέλφων και του κύριου Χάστινγκ. ότι περί ότι υπονομεύεται ε, ο περιορισμός των ε, μέτρων στην χρήση τους ως προς το σκοπό και η πρόσβαση στη Eurodac ήταν τελείως διαφορετική, υπό τελείως διαφορετικές προϋποθέσεις όταν θεσπίστηκε. Το δικό μας μέλημα και η ανησυχία που διαρκώς εντείνεται είναι ακριβώς αυτή, ότι ποιος ε, θα εμποδίσει. Ανα πάσα στιγμή υπάρχει ένας κατάλογος ή μια βάση δεδομένων να έρθουν οι αρχές και να πούνε χρειαζόμαστε πρόσβαση. Και εκεί αρχίζει βέβαια άλλη συζήτηση τελείως διαφορετική από αυτήν που είχε γίνει όταν θεσπίστηκε η βάση δεδομένων. Και γι' αυτό θέλουμε αυστηρή τήρηση της αρχής της αναλογικότητας. Συμφωνώ με τον κύριο Χαστίν, δεν είναι τεχνικού χαρακτήρα το εγχείρημα. Δεν μπορούμε να έχουμε προσέγγιση με την οτροπία του Δούνε και λαβίνα του έναντι για κάποιο άλλο μέτρο στο πακέτο του ασύλου. Και κλείνοντας θεωρώ ότι είναι πολύ δυστυχής η επιλογή της πρόσβασης των δεκτικών αρχών σε μια βάση δεδομένων για το άσυλο, πράγμα το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από το μέτρο που εγώ είχα διαπραγματευτεί με το Συμβούλιο, τη δυνατότητα πρόσβασης δηλαδή στην βάση δεδομένων δις όπου είναι επισκέπτες, είναι άνθρωποι οποίοι έχουν επιλέξει να έρθουν σε μια χώρα και έτσι είναι διαφορετική η χρήση. Αυτό που δεν καταλαβαίνω επακριβώς είναι τι είδου μέτρα μπορεί να εισαχθούν εάν ε, παραδείγματι επιτύχουν στον εντοπισμό κάποιου από τα δακτυλικά αποτυπώματα οι αρχές. Θα είναι του, η, ε, η, η απόφαση του 2006 960 σε εφαρμογή εφόσον υπάρχει μια ταυτοποίηση. Και εφόσον υπάρχει ταυτοποίηση και αρχίσει μια ανακριτική διαδικασία, τι γίνεται με την τιμή, τι θα έχει το άσυλο στο μεσοδιάστημα, γιατί δεν λέγεται τίποτα γι' αυτό. Για το άρθρο 211 ε, για τα δακτυλικά αποτυπώματα, τα λεγόμενα λανθάνοντα latent, εννοείται μερικά αποτυπώματα από λανθάνοντα που έχουν συλλεγεί σε, μία, ε, σε ένα τόπο εγκλήματος. Υπάρχει ζήτημα αξιοπιστίας εδώ. Λανθάνοντα αποτυπώματα που συλλέγονται από τόπο εγκλήματος. Μερικά μπορούν πράγματι να ταυτιστούν από τη βάση δεδομένων της Eurodac. Υπάρχουν κάποιες προβλέψεις με ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Επίσης, στα όσα είπε ο κύριος Χάστινγκς για το ρόλο ή τη φύση της αρχής επαλήθευσης του άρθρου 6. Θα είναι ανεξάρτητη, τι είδους αρχή θα είναι αυτή, θα έχει δικαστικό χαρακτήρα, όλα αυτά προς το παρόν. Το κείμενο του Συμβουλίου τα αφήνει να τα κρίνουν τα κράτη-μέλη. Θα ήταν καλό να είχαμε πιο συγκεκριμένα κριτήρια στην επιλογή της εν λόγω αρχής. Επίσης υπάρχει η αποτυχία συλλογής ε, καταγραφής τακτικών αποτυπωμάτων από έναν ετούντα στο κείμενο, στην πρόταση, ε, αντιμετωπίζεται μόνο το ενδεχόμενο μιας προσωρινής αποτυχίας. Εάν είναι μόνιμη η αποτυχία της ε, συλλογής δακτυλικών αποτυπωμάτων, δεν θα πρέπει να πάμε στην άλλη λύση που ισχύει για το βρύς. Επίσης, μια παρέκκληση για ε, έκτακτες περιπτώσεις κατεπήγοντος που προτείνει να μην γίνεται επαλήθευση εάν πράγματι υπάρχει αυτή η επίγουσα ανάγκη και η άνευ αδικαιολογή του καθυστερήσεως αναφορά. Πάλι δεν είναι σαφής για μένα χωρίς να μπορώ να παραθέσω το επακριβές κείμενο της ε, εν λόγω αποφάσεως του 2006, θα ήθελα να δω εάν πράγματι υπάρχει αντίστοιχη αναφορά στο κείμενο της αποφάσεως του 2006. Στο άρθρο 20 και τις προϋποθέσεις πρόσβασης στη Eurodac των αστυνομικών αρχών δεν αναφέρεται τίποτα. Δεν ορίζονται πουθενά παράμετροι υποχρεώσεων ε, για ένα κράτος μέλος. Να πρέπει δηλαδή να επαληθεύει άλλες εθνικές βάσεις δεδομένων ε, με κάποιο άλλο τρόπο. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιες άλλες εναλλακτικές πριν φτάσει στην ε, Eurodac το κράτος μέλος, Εκτικές αρχές. Δεν θα πρέπει πρώτα να περάσει περίπου από τη ΒΙΣ. Επίσης, ε, στο κείμενο του Συμβουλίου έχει απαλληφθεί το κριτήριο ότι, ότι πρέπει να υπάρχουν επαρκείς λόγοι που να επιτρέπουν το συμπέρασμα ότι χάρη στη βάση δεδομένων Eurodac μπορεί να αποτραπεί να διαλευκανθεί ένα, ένα έγκλημα. Μπορεί να διαλευκανθεί συγγνώμη ένα έγκλημα κτλ. Δηλαδή ούτε καν η προϋπόθεση της εύλογης απόδοσης μιας ε, επιτυχίας, εύλογης πιθανολόγηση της επιτυχίας της έρευνας. Όχι απόδειξη επιτυχίας, αλλά πιθανολόγηση. Ούτε καν αυτό δεν προβλέπεται. Ακόμη και εδώ λοιπόν το κριτήριο αυτό που ήταν μάλλον ασθενές έχει απαλληφθεί από το Συμβούλιο. Στο άρθρο 21 δεν προβλέπονται κριτήρια για την πρόσβαση στη της Europol, άμεση ή έμεση, φερειπίν το EDPS. Θα πρέπει να εξετάζει τα αιτήματα της Europol, θα ήταν εφικτό κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, αλλά πάλι θα επιμένω ότι θα πρέπει πάντα να επαληθεύουμε ότι ισχύουν ε, τα, ε, τα κριτήρια και οι προποθέσει. Συνεχίζω και τελειώνω, Πρόεδρε, με το άρθρο 29 που αναφέρει ότι θα πρέπει ο ετών το άσυλο να ενημερώνεται μόνο για τους στόχους του κανονισμού του Δουβλίνου και ότι δεν υπάρχει κανένας ε, λόγος να ενημερωθεί από τις αστυνομικές αρχές ότι μπορεί να έχουν ε, πρόσβαση στα δακτυλικά του αποτυπώματα ή να ενημερωθεί ο ετών ότι μπορεί να δοθεί η πρόσβαση στι αστυνομικε αρχε στα αποτυπώματά του. Εδώ πάλι βλέπω κενό. Στο 234 όπου αναφέρεται ότι μπορεί να απαλληφθεί εάν δεν εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη ε, ανακριτική διαδικασία. Αλλά το υλικό της Eurodac αναφέρεται ότι θα πρέπει να είναι ε, χρήσιμο, απαραίτητο, σε μια συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν το 33-4 τι θέλει. Μόνο για συγκεκριμένη υπόθεση μπορεί να το ζητήσει. Άρα προφανώς και θα πρέπει να απαλληφθεί εάν δεν χρειάζεται πλέον σε μια συγκεκριμένη υπόθεση. Τι σημαίνει αυτή η χωριστή αναφορά. Θα διαγράφεται το υλικό εάν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα για την οποία να έχει χρησιμοποιηθεί ή μπορεί να διακρατηθεί από την αστυνομία και να χρησιμοποιήσει σε άλλη ενερεξελίξη ενδεχομένω ε, έρευνα. Αυτά, ζητώ συγγνώμη που επέμπεινα σε αυτές τις λεπτομέρειες, είναι σημαντικές όμως και δεν ξέρω αν ε, θα μπορούσε έστω η Επιτροπή παραδείγμα να μου δώσει γραπτός μια απάντηση, αν θεωρώ ότι δεν μπορεί να απαντήσει σήμερα στις ερωτήσεις αυτές. Θεωρώ πάντως ότι πρέπει να είμαστε πολύ, πολύ προσεκτικοί στην εξέταση αυτών των μέτρων. Και αυτό εξηγεί και τι καθυστερήσει. Δεν έχουμε προχωρήσει στο θέμα του Ιουροτακό όσο γρήγορα θα θέλαμε εμεί στην Επιτροπή μα. Αλλά πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί, πρέπει να επαληθεύεται σε κάθε σημείο η συμβατότητα αυτού του μέτρου που επιτρέπει την ε, πρόσβαση στι αστυνομικέ αρχέ τη βάση δεδομένων. Εγώ δεν ε, είμαι αφελή, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν ενδεχομένω εγκληματίε μεταξύ αυτών που καταθέτουν έτσι για άσυλο. Αλλά βασική αρχή το τεκμήριο της αθωότητας και ως εκ τούτου στοιχεία τα οποία συλλέγονται για ένα συγκεκριμένο σκοπό δεν νομίζω ότι μπορούμε να λέμε ότι αν εφετέρου θα έχει πρόσβαση η αστυνομία σε αυτά. Και δεν νομίζω ότι μπορούμε να το θεωρήσουμε και σε μια βάση μια συγκεκριμένη πολιτική ε, συμφωνία διαπραγματεύση. Ευχαριστώ πολύ. Πριν στραφώ στην Επιτροπή έτσι ώστε να απαντήσει στα ερωτήματα που ετέθησαν, θα ήθελα και εγώ να θέσω δύο ερωτήματα εξ ονόματος του συναδέλφου Κλοντ Μωράες, ο οποίος ε, αναγκάστηκε να φύγει. Δύο ερωτήματα προς την Κομισιόν λοιπόν. Πρώτον, το Συμβούλιο και η Κομισιόν τι λένε όσον αφορά την ε, ε, ε, όσον αφορά την θέση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την προστασία προσωπικών δεδομένων ότι δεν υπάρχει αναλογικότητα. Επίσης, μπορεί να μας εξηγήσει η Κομισιόν γιατί η γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Εποπτείας δεν ζητήθηκε εκ των προτέρων. Αυτά τα δύο ε, ερωτήματα, τα οποία θα προσθεθούν βέβαια στα ερωτήματα που έθεσαν προς την Κομισιόν και μετά θα επανέλθουμε ε, στον εισηγητή μας. Η Κομισιόν παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κατανοείτε φαντάζομαι ότι δεν μπορώ να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις, αλλά θα προσπαθήσω να απαντήσω στα πιο σημαντικά σημεία. Και βεβαίως είμαστε στη διάθεση των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για περαιτέρω συζήτηση των θεμάτων. και έτσι ώστε να λυθούν παρεξηγήσεις ε, οι οποίες ε, θα επιτρέψουν εν τέλει την λύση των ε, προβλημάτων αυτών. Να πω καταρχάς ότι η Κομισιόν λαμβάνει υπόψη όλα τα όσα αναφέρει η συγγήτρια στην έκθεσή της. Το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και σε σχέση και με την ε, μελέτη επιπτώσεων ε, πρέπει να πω, το είπα και την προηγούμενη φορά, ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι απολύτως παρόμοια με την πρόταση του 2009 για την πρόσβαση στο, του στο σύστημα Eurodac από τις αρχές επιβολής του νόμου λαμβάνονται υπόψη όσο γίνεται περισσότερο και οι προτάσεις του Συμβουλίου όπως γίνεται και αυτή τη στιγμή λαμβάνοντα υπόψη τη νέα πρόταση της Κομισιόν είναι παρόμοια προ την ε, πρόταση του 2009, κατά την άποψή μα, ε, η ίδια μελέτη επιπτώσεων μπορεί να ισχύσει και επομένως κατά την άποψη της ε, Κομισιόν δεν υπήρχε λόγο για νέα μελέτη επιπτώσεων και με όλο το σεβασμό δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει το πολιτικό τοπίο, η θέση ισχύ της συνθήκης Λισαβόνας κατά την έννοια αυτή. Επιτρέψτε μου επίσης να ασχοληθώ με το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Υπάρχουν σημαντικές επιπλέον πληροφορίες στο κεφάλαιο 3 Εκεί μελετάται η επίπτωση της πρότασης ε, κυρίως στη διαδικασία αιτήσεως ε, ασύλου και την προστασία προσωπικών δεδικαιωμένων ε, και ε, ε, υπάρχει πλήρης ε, ευθυγράμμιση και σεβασμός του αντιστοίχου κεφαλαίου το, της, του χάρτας των θεμελιδών δικαιωμάτων και ταυτίζεται επίσης και με το κεφάλαιο 3 του επεξηγηματικού μνημονίου. υπομνήματος συγγνώμη. Όσον αφορά το EDPS, η Κομισιόν είναι ανοιχτή σε προτάσεις και συστάσεις. Πρέπει να πω ότι και η συζήτηση στο Συμβούλιο έχει καταδείξει ότι ε, θα πρέπει να ε, υπάρξει ε, σαφής διαχωρισμός στην δυνατότητα χρήσης των δακτυλικών αποτυπωμάτων βάσει του συστήματο Eurodac. Επίση, μπορεί να συμφωνήσει η Κομισιόν ότι τη στιγμή που λαμβάνονται τα δακτυλικά αποτυπώματα θα πρέπει να υπάρξει ε, και η απαραίτητη ενημέρωση ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα αποτυπώματα αυτά για θέματα επιβολής νόμου και ότι ε, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει οπωσδήποτε ε, να ασχολείται με το θέμα αυτό εμπειρογνώμων των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Επίσης, να επαναλάβω αυτό που είπα και στην τελευταία μας ε, συνάντηση, στην παρουσίαση της προτάσεως της Επιτροπής η πιστεύει ότι η πρόταση είναι ε, αναλογική, ε, παρουσιάζει πολλά καλά στοιχεία, και ε, είναι γεγονός ότι ο έλεγχος μέσω του συστήματος Eurodac θα είναι πραγματικά η τελευταία, ε, το τελευταίο σημείο, η τελευταία προσφυγή που θα έχει κανείς. Καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό πολιτικό ε, ζήτημα αλλά ε, ε, ε, οφείλω να πω, όπως το έχω ξαναπεί, ότι θα χρησιμοποιηθεί μονάχα σαν ίστατο εργαλείο και μονάχα για ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήματα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να, για συστηματική χρήση ή συστηματική πρόσβαση του συστήματος Eurodac, ούτε υπάρχει δυνατότητα και πιθανότητα μεταβίβασης των στοιχείων σε άλλες χώρες. Θα να ασχοληθώ τώρα σε κάποια από τα ερωτήματα τα οποία έθιξαν, ε, ε υπέβαλαν μάλλον οι βουλευτές. Η κυρία Κέλλερ ε, δεν ε, υπάρχει, λέει, απαραίτητη επεξήγηση όσον αφορά την δυνατότητα χρήσης του συστήματος Eurodac από την Europol. Να σας πω δύο-τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα η Europol αποτελεί ένα κόμβο πληροφοριών για την Ευρωπαϊκή Ένωση. και γι' αυτό πιστεύουμε ότι και η Europol θα πρέπει να έχει πρόσβαση. Δεύτερο λόγο είναι ότι η Europol παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε την ε, καταπολέμηση του τράφικινγκ ε, και επομένως με τον τρόπο αυτό μπορεί να προστατέψει θύματα του τράφικινγκ, θύματα ε, της εκμετάλλευσης και μπορεί να αποτρέψει την, ε, ε, το τράφικινγκ. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύουμε ότι θα πρέπει να έχει πρόσβαση στο σύστημα Eurodac Europol και αυτό ε, το έχω ξαναπεί. Φυσικά οι ετούντες άσυλο είναι ευάλωτη ομάδα και αυτό μάλιστα κατεδείχθη και στην ε, μελέτη επιπτώσεων ε, του 2009. Επομένως ε, θέλουμε να τους προστατέψουμε και δεν θέλουμε προστασία αυτή να δυναμητιστεί από την πρόταση αυτή. Όπως και στο επεξηγηματικό υπόμνημα αναφέρουμε, πιστεύουμε ότι είναι ε, ε, θα, θα πρέπει να αποτραπεί οποιοδήποτε στιγματισμός των ετούντων άσυλο λόγω αυτής της δυνατότητας πρόσβασης στο σύστημα Eurodac. Ε, επ' αυτού θα, μελετηθεί, επ θα μελετήσουμε το ζήτημα και θα επανέλθουμε. Η Βαρονές Λάτφορτ αναφέρθηκε στην ανεξαρτησία της ε, ε, ελεγκτικής αρχής αυτό είναι όντως αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο κατανοεί το θέμα η Κομισιόν δηλαδή ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, ευλήρης ανεξαρτησία των αρχών η, η αρχή ελέγχου και η αρχή διακρύβωσης θα πρέπει να είναι απολύτως ανεξάρτητες. αλλά εάν χρειάζονται περαιτέρω αφηνήσεις, μπορούμε να το συζητήσουμε διμερώς μαζί σας. Ένα άλλο σημείο το οποίο θίγει είναι ότι η ε, μελέτη επιπτώσεων της ε, Κομισιόν δεν έδειξε την ε, αναλογικότητα της χρήσης για την επιβολή του νόμου. Βεβαίως αυτό είναι ένα νέο εργαλείο, είναι δύσκολο να πούμε κάτι τέτοιο, αλλά όπως είπα και στην τελευταία μας συνάντηση, Κατά την ε, άποψή μας η πρόταση έχει, ε, μάλλον κλείνει ένα κενό ε, δομικό Γιατί με τον τρόπο αυτό μπορεί κανείς να βρει στοιχεία τα οποία δεν βρίσκονται ούτε στα στοιχεία πριν. Επίσης, Σήμερα πρέπει να σας πω ότι ήδη είναι δυνατόν να ανταλλαγούν στοιχεία ε, ετούντων άσυλο μεταξύ των ε, κρατών μελών, ε, βεβαίως υπό το ενωσιακό καθεστώς, υπό την ενωσιακή νομοθεσία. Έχουμε κάποιες, έχουμε παραδείγματα της χρήσης. Α, μας ζητάτε, παραδείγματα ε, για το κατά πόσον έχει βοηθήσει η προσφυγή στο σύστημα Eurodac για την καταπολέμηση οργανωμένου εγκλήματος. Μα μέχρι τώρα δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο, άρα δεν έχουμε παραδείγματα. Η Βαρονέσα Λάτφορτ ε, έθεσε ένα ερώτημα σχετικά με τις ε, περιπτώσεις όπου υπάρχει hit ε, στο εθνικό σύστημα. Ε, αυτό σημαίνει ότι η περαιτέρω αντιμετώπιση των δακτυλικών αποτυπωμάτων θα γίνει σε εθνικό επίπεδο μέσω των εθνικών διεργασιών. Και επίσης ε, ρώτησε η ίδια βουλευτής εάν μερικό αποτύπωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ναι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Όμως, και εδώ Έχουμε ίδια άποψη με την εισηγήτρια του EDPS. Ε, θα πρέπει στην στο πρώτο αίτημα να υπάρχει hit. Εάν είναι no hit, τότε αυτό σημαίνει ότι ε, είτε δεν υπάρχει τίποτα, είτε η ποιότητα δεν ήταν ικανή για να υπάρξει hit. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι από τη δική μου πλευρά τουλάχιστον έχω, κατα... έχω ε, καλύψει ε, τα περισσότερα ε, σημεία και βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λάτφορτ, χωρίς μικρόφωνο. Ναι, μια συμπληρωματική ερώτηση πολύ σύντομα για την Επιτροπή γιατί δεν ξέρω πως φταίω εγώ και δεν κατάλαβα το όλη τη βδομάδα έχω κουραστεί. Μου είπατε ότι ήδη ναι. έχουν προβεί σε ανταλλαγή στοιχείων από τη Eurodac για λόγους ναι. επιβολής του νόμου τα κράτη-μέλη μεταξύ τους. Αυτό δεν επιτρέπεται, έτσι δεν είναι. Δηλαδή αν έχουν αρχίσει να προβαίνουν σε αυτές τις ανταλλαγές, ενώ δεν επιτρέπεται, γιατί το κάνουν ή γιατί τους αφήνεται να το κάνουν. Όχι, όχι, Βαρόνι Λάτφορτ, υπάρχει μια παρεξήγηση τα κράτη-μέλη ανταλλάσσουν εθνικά δεδομένα. Εθνικά δεδομένα μπορούν να ανταλλάσσουν. Εθνικά δεδομένα τα οποία καταγράφουν από ετούντε στο άσυλο. Με τη διαδικασία. Η Eurodac απλώς απλουστεύεται αυτή η διαδικασία. Ένα που φτάνει στο Ηνωμένο Βασίλειο για να στήσει άσυλο, μπορεί να καταθέσει, παίρνουν, τα αποτυπώματα και μπορούν τα αποτυπώματα αυτά να τα διαθέσουν στα άλλα κράτη-μέλη για του στοχού τη. Δηλαδή, βασικά και τη βήτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο, μα λέτε, λέει η κυρία Λάτφορτ. Θέλετε μήπω και εσεί να μα δώσετε κάποια συμπεράσματα. Κύριε Φω, εσεί. Η Προεδρία. Η Προεδρία θέλει να πει παρακαλώ κάτι εκ μέρου τη Κύπρου. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Φυσικά είναι δύσκολο, όπως αντιλαμβάνεστε για μένα, να συνοψίσω όλα τα όσα ακούστηκαν και να υποθέσω αυτά που θα ήθελε να πει η, ε, η συγγήτρια. Πάντως από τη συζήτηση μπορώ να πω συνοπτικά ότι τα θέματα αυτά τα οποία έχουν μια σημασία μεγάλη αλλά μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική αποδοχή πιστεύω είναι σημεία στα οποία θα πρέπει να επιμείνουμε, να τα επεξεργαστούμε, να τα διατυπώσουμε σε τροπολογίες και βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη τις τοποθετήσεις που ακούστηκαν. Εν γέννη, το θέμα δεν είναι μόνο ε, να εξασφαλιστεί μια δομή μέσα στην Ευρώπη για το τόσο σημαντικό δίκαιο του ασύλου, αλλά και να υπάρχει κατάλληλη διαδικασία για αυτό. Και έτσι εδώ έχουμε τα διάφορα επιμέρους προβλήματα που θα πρέπει να εξεταστούν, όπως άλλωστε μας εξήγησε και ο κύριος Χάστινγκς. Είπαμε, σκοπιμότητα, πρόσβαση εθνικών αρχών, η οποία θα πρέπει μόνο και σε ε, κατά περίπτωση εξεταζόμενες προϋποθέσεις ε, ιδιαίτερη ανάγκης και με αυστηρούς όρους να έχουν πρόσβαση στις βάσεις, στη βάση δεδομένων. Και η σκοπιμότητα αυτή λοιπόν που αναφέρω θα πρέπει ταυτόχρονα να, επισημε... να αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από άλλα μέτρα για την τήρηση της ασφάλειας. Πρέπει να υπάρχουν τεσφαλιστικές δικλείδες για τον τρόπο με τον οποίο θα ε, χειριστεί τα στοιχεία αυτά η ιδιοκτική αρχή. Όπως πολύ σωστά επεσήμανε και ο κύριος Χάστινγκς, αν και σημειώνω τις παρατηρήσεις του για την εποπτεία από μια ανεξάρτητη αρχή και την χρήση με βάση τον στόχο για τον οποίο έχουν συλλεγεί τα στοιχεία, τη σκοπιμότητα δηλαδή. Και στην ε, συνεδρία των σκιωδών συγγητών ασφαλώς θα τα εκθέσουμε και θα τα συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Κύριε Φως, που εκπροσωπείτε την κυρία Μακοβέη. Ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες, τον κύριο Χάστινγκς φυσικά, που έλαβε μέρος στην πολύ ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση και ήρθε η ώρα να σα ανακοινώσω προθεσμία για τις τροπολογίες 7 Νοεμβρίου, 7 Νοεμβρίου, κατάθεση τροπολογιών, εξέταση του 26-27 Νοεμβρίου, ψηφοφορία ανατολισμου 17-18 Δεκεμβρίου, όπως σήμερα απεφάσισαν οι συντονιστές και σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Περνάω στο επόμενο θέμα, το υπαριθμό 15. Ευχαριστώ in this long day. There goes. So, if you don't mind, we move on to point number 15, which is asylum. Άσυλο. Άρθρο 15, Ταμείο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση. Κυρία Γκυλιόμ, θα μας κάνει την παρουσίαση. τις προτάσεις των τροπολογιών και μετά θα ακούσουμε Επιτροπή, Συμβούλου κτλ. Κύριε Αγγίωμ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, γρήγορα όσο πιο γρήγορα είναι δυνατό. Μερικά σχόλια για τις τροπολογίες που κατατέθηκαν για αυτήν την έκθεση είναι 120. Πολλές ε, έχουν εκεί, συνυπογράφονται από τα μέλη. Και αυτό είναι καλό κατά τη γνώμη μου. Ένα άλλο πράγμα που βρίσκω θετικό είναι ότι και τις τροπολογίες τις δέχομαι θετικά διότι εντάσσονται στη γενικότερη γραμμή της έκθεσης και υποστηρίζουν την πρόταση της Κομισιόν ενισχύοντας ορισμένες διατάξεις ή διευκρινίζοντάς τις. Για να σας αναφέρω στα γρήγορα το πακέτο των τροπολογιών που κατατέθηκε, οι στόχοι που προσπίζονται είναι οι εξής. Υπογραμμίζουν τη σημασία της τεχνικής βοήθειας, είναι σαφές ότι η διάρθρωση και η εσωτερική λειτουργία έχουν απλωστευτεί, οπότε και το διοικητικό κόστος θα είναι ε, πιο ελαφρύ για τα κράτη-μέλη, αλλά τα κράτη φυσικά πρέπει να υποστηριχθούν για να χρησιμοποιήσουν, να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο αυτά τα κονδύλια. Καλούνται επίσης τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν την διαφάνεια ε, και να θέσουν σε εφαρμογή άμεσα το Ταμείο. Επίσης, να έχουμε μία δίκαιη και διαφανή χρήση των ε, πιστώσεων. Είναι πολύ καλό πράγμα όλο αυτό το θέμα της ε, κατανομής ε, της χρηματοδότησης για τις τρεις προτεραιότητες, για το υποδοχή, άσυλο κλπ. Και δεν θα πρέπει να ευνοήσουμε τη μία επιλογή ε, στο άλλο, δηλαδή να έχουμε μία προσέγγιση καθαρά ασφάλειας ε, που και να επιβαρύνει την ε, πλευρά ανθρώπινη προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το άλλο πακέτο αφορά στην πλαισίωση και τη χρηματοδότηση των οργανισμών της Ένωσης μέσω του Ταμείου για το Άσυλο και τη Μετανάστευση. Δεν αμφισβητώ καθόλου ότι αυτή η χρηματοδότηση θα μπορούσε να πάει προς τους οργανισμούς, αλλά δεν θα πρέπει όμως αυτά τα ταμεία να χρησιμοποιηθούν ως ένα μέσο για να καλύψουν τρύπες στον προπολογισμό των οργανισμών. Και έχω κατά νου δηλαδή ότι πρέπει να παρακολουθούμε από κοντά τη χρηματοδότηση του Frontex, γιατί ο κύριος Λαϊτίνεν σήμερα το πρωί μας είπε ότι θα πάει να ψάξει χρήματα αλλού. Τώρα, έχω άλλα ε, έχω και άλλες ε, τροπολογίες. Έχουμε λοιπόν ε, και το θέμα της ενίσχυσης της ποιότητας σχετικά με την επανεγκατάσταση. Έχω καταθέσει ένα σωρό τροπολογίες για αυτό το θέμα. Για τις άλλες ε, τροπολογίες επιμένω για, τις, ε, για τρεις ε, διαστάσεις υπάρχει ένα σαφώς μήνυμα που έστειλε το Κοινοβούλιο σχετικά με την αλληλεγγύη. Όλοι θελήσαμε να καταθέσουμε μία τροπολογία έχοντας το άρθρο 80 ως νομική βάση πρόκειται για ένα ισχυρό μήνυμα και το οποίο λέει ότι όλο το Κοινοβούλιο ασχέτως πολιτικών προσανατολισμών είναι ενωμένο και θέλει να περάσει ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Το δεύτερο τμήμα πάλι αφορά στην ανάλυση για την καλύτερη χρήση των κονδυλίων και ανάλυση και των χρηματοδοτούμενων, χρηματοδοτούμενων δράσεων, ε, επίσης ε, κατανομή και για το ποσοτικό σκέλος και το ποιοτικό σκέλος, καλύτερη διαβίβαση πληροφοριών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε αυτή τη διάσταση μου φάνηκε να κατάλαβα ότι το Συμβούλιο θα υποβάλει μία πρόταση να μπουν όλες αυτές οι διατάξεις στο παράρτημα. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αποφασίσουμε. Αλλά η αξιολόγηση και ανάλυση του ρίσκου είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Τώρα ένα ποιοτικό και ποσοτικό άλμα για τα θέματα επανεγκατάστασης. Πολλές τροπολογίες έχουν κατατεθεί σχετικά και αυτό αποδεικνύει ότι το Κοινοβούλιο θέλει να εκφράσει μία Ευρώπη ασύλου και αλληλεγγύης. Ο κύριος Σταβάρης και εγώ έχουμε καταθέσει από κοινού τροπολογίες οι οποίες λένε ότι πρέπει να κάνουμε, να πράξουμε καλύτερα και να κάνουμε περισσότερα. Δηλαδή το ποιοτικό και το ποσοτικό σκέλος. Επίσης, εξαγγελία προγραμμάτων επανεγκατάστασης και να έχουμε μία ποιοτική προσέγγιση για την ποιότητα ή υποδοχής και την ποιότητα της, ε, ε, την ευημερία των, ε, των ανθρώπων που, έχουμε επανεγκαταστήσει. Αυτά κύριε Πρόεδρε, θα έχουμε ε, το Νοέμβριο μία ψήφο με προσανατολιστικό χαρακτήρα και εγώ θα κοιτάξω να μαζέψω και τους στιώδεις εισηγητές για να κοιτάξουμε να βρούμε λύσεις για τους συμβιβασμούς. Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Καιρό είναι τώρα να ακούσαμε το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Έχετε το λόγο σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε την εισηγήτρια, καθώς επίσης ε, και τους βουλευτές ε, που υπέβαλαν τροπολογίες. Να σας πω καταρχήν ότι το Ταμείο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση είναι ε, μέρος της δέσμης ε, για το πακέτο των ε, προοπτικών και τα άλλα δύο εργαλεία θα είναι το Ταμείο της Εσωτερικής Ασφάλειας θα συζητηθούν στην επόμενη συνεδρίαση της Λιμπεάν, κατάλαβα καλά θα ασχοληθώ με τα γενικά σημεία τα οποία αφορούν την έκθεση και τις τροπολογίες, αλλά μπορούν να ισχύσουν και για, τις, για τα άλλα ταμεία. Ε, πρώτον, ε, θεμελιώδη δικαιώματα. Βεβαίως, συμμερίζεται η Κομισιόν την σημασία που αποδίδει το Κοινοβούλιο στο θέμα αυτό. Καμία πρόθεση ουδέποτε είχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μειώσει την δυνατότητα πολιτών τρίτων χωρών να ε, υποβάλουν αίτημα ασύλου. Και βεβαίω η συμμόρφωση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλες αρχές ε, ε, είναι άρρητα συνδεδεμένε με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου και θα στηριχτούν περαιτέρω από το Μείο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση. Υπάρχουν τροπολογίε σε διάφορα άρθρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και ενδεχομένω εδώ μπορούμε να συζητήσουμε ε, για να μπορέσουμε να βρούμε ε, εξ αρχή κάποιου κάποιους Γιατί ε, είναι μια αρχή η οποία εφαρμόζεται σε όλο το κείμενο. Οι δείκτε τώρα που ανέφερε και η συγχύτρια όπως είπα και την τελευταία φορά που ήρθα να μιλήσω στην Επιτροπή Λίμπε για το εργαλείο αυτό, οι δείκτες οι οποίοι αναφέρονται στο κείμενο είναι ενδεικτικοί. Είχαμε συμφωνήσει με τα κράτη-μέλη και το είπαμε και στο Κοινοβούλιο, ότι θα συζητήσουμε κοινού δείκτες στα εργαστήρια και επί τη βάση αυτού της, της η Προεδρία θα υποβάλει νέο κείμενο προς συζήτηση στο Συμβούλιο. Την προηγούμενη εβδομάδα έγιναν αυτά τα εργαστήρια και ήταν μάλιστα καλεσμένο και το Κοινοβούλιο και ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει ε, συζήτηση την επόμενη εβδομάδα στην Ad Hoc Επιτροπή του Συμβουλίου και βεβαίως ε, συζητήθηκαν και οι τροπολογίες που έχουν υποβληθεί από την Επιτροπή σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να παραμείνουν οι δείκτες ε, ε, πολύ απλοί. Να θυμίσουμε ότι οι δείκτες που αναφέρονται στο κείμενο είναι κοινοί δείκτες. Συνδέονται με την ειδική σκοπιμότητα του Ταμείου και πρέπει να αντικατοπτρίζουν, να είναι σε θέση να αντικατοπτρίζουν την στήριξη που δίνεται σε συγκεκριμένους τομείς από το Ταμείο που, ή που πρέπει να καλύπτονται από το Ταμείο. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει κάθε χρόνο να κάνουν αναφορά ε, βάση, ε, σε αιτήσια βάση και μάλιστα βάση αυτών των προβλεπόμενων δικτών. Προβλέπονται επίσης και κάποιοι ειδικοί δείκτες, συζητήθηκε και αυτό στο, στην ομάδα εργασία. Αλλά οι κοινοί δείκτες ε, θα πρέπει, οι κοινοί γενικοί δείκτες θα πρέπει να είναι απλοί και εύχρηστη. Ένα άλλο σημείο στο οποίο αναφέρθηκε η συγγήτρια είναι η τεχνική αρρωγή. Βεβαίω η τεχνική αρρωγή είναι σημαντική. και έχουμε τεχνική αρρωγή και στο ε, μελλοντικό ταμείο 5% για τεχνική ε, αρρωγή που είναι παραπάνω από την πρόταση για τα ε, διαρθρωτικά ταμεία και ξεπερνάει και το παρόν ε, ποσοστό που είναι 4,3%. We fully explain the situation on technical assistance. Για το Ταμείο Αλληλεγγύης η συζήτηση στο Συμβούλιο για αυτό και για τα άλλα, στην συζήτηση μάλλον, ε, και για αυτό και για άλλο ταμείο προβλέπονται ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες θα έχουν μικρότερα προγράμματα και το πάγιο κόστος ε, και τα χρήματα τα οποία θα ε, πάρουν για την τεχνική ε, στήριξη δεν θα είναι αρκετά. Πάντως απεφασίσει ότι τα κράτη-μέλη ανεξαρτήτως πόσο μικρό είναι το πρόγραμμα θα έχουν ένα σταθερό ποσό τεχνικής αρρωγής. Όμως το 7% είναι πάρα πολύ ε, μεγάλο για την Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή και ε, πρέπει να πούμε ότι όσο περισσότερα κονδύλια δαπανώνται για τεχνική αρρωγή, τόσο λιγότερα χρήματα μένουν για την πραγματική δράση επιτόπου. Καλύτερα λοιπόν είναι να υπάρχουν περισσότερα κονδύλια διαθέσιμα για τις ε, πραγματικές διαδικασίες, ε, για τις πραγματικές πανεμβάσεις ε, από τις οποίες θα ωφεληθούν τελικά οι δικαιούχοι. Επίσης, να πω ότι όλες οι υπηρεσίες ε, έχουν ένα ε, ε, επίδομα από, τις, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βάσει των πολιετών βάλει του πολιετού πλαισίου και όπως άλλωστε αναφέρεται και στο επεξηγηματικό υπόμνημα, θα μπορούσαμε να προβλέπουμε σε εξαιρετικές συνθήκες να ε, δοθούν κάποιες ad hoc επιπλέον αρμοδιότητες στις υπηρεσίες ε, ε, κατά παράβαση, κατά εξαίρεση μάλλον, του δημοσιονομικού κανονισμού. Αυτά τα, αυτό το ταμείο για το άσυλο και την μετανάστευση και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας δεν είναι δευτερογενής πηγή χρηματοδότησης και επομένως δεν μπορεί να δεχτεί η Κομισιόν τις τροπολογίες 174 και 184. Αν μου δώσετε λίγο χρόνο ακόμα θα μπορούσα να σχολιάσω κάποιες από τις τροπολογίες οι οποίες είναι πάρα πολύ ε, συγκεκριμένες για το άρθρο 80, επί του οποίου η εισηγήτρια αναφέρθηκε. Η άποψη της Κομισιόν είναι ότι η νομική βάση την οποία έχουμε επιλέξει είναι ικανή. Όμως αναγνωρίζουμε Ε, και βάσει της ανακοίνωσης ε, του Μαρτίου του 2012 είμαστε έτοιμοι να το ξανασκεφτούμε υπό το φως και των σχολείων που έκανε η εισηγήτρια. Δεύτερο, ε, οι ομάδες στόχοι. Η τροπολογία 121 αναφέρει ότι ένα, ε, ε, μια ομάδα στόχος θα μπορούσε να είναι ε, αυτοί οι οποίοι διαμένουν σε άλλη χώρα. Οι, πολίτες, οι Ευρωπαίοι πολίτες οι οποίοι ζουν σε άλλες χώρες απλώς ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης που έχουν και επομένως δεν μπορούν να μπουν στο MFF. για το άσυλο η τροπολογία 102 προτείνει ένας νέος ειδικό στόχος να προσθεθεί έτσι ώστε να στηριχτούν ε, μέτρα ε, για την ε, σωστή πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου. Νομίζουμε ότι υπάρχει ήδη ένα κεφάλαιο το οποίο αφορά την ενδυνάμωση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Εκεί εμπίπτει αυτό. Πάντω, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για την επικοδομητική στάση και τις επικοδομητικέ τροπολογίες. Η εισηγήτρια ανέφερε την σημασία του να δοθούν, ε, τη, συγγνώμη, τη σημασία της κινητροδότησης, έτσι ώστε τα, τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν και νέα κίνητρα. Ε, μας ενδιαφέρει να αυξήσουμε την δυνατότητα ε, των ε, ετούντων ασυλών να δουν την κατάστασή τους να σταθεροποιείται. Αυτό μας βρίσκει σύμφωνος, αλλά δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με ένα καταπολύπη ποσό το οποίο θα δίνεται σε όλους. Θα πρέπει επίσης να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε την προσπάθεια απλούστευσης, κύριε Πρόεδρε. Ε, τα κράτη-μέλη ε, έχουν ε, ήδη την δυνατότητα να δαπανίσουν τους πόρους τους για την οικοδόμηση ικανότητας. Επομένως, κατά την άποψή μας, δεν, νομίζω ότι υπάρχει, δεν νομίζουμε ότι υπάρχει λόγος να ληφθούν οι υπόψη περαιτέρω στόχοι και μάλιστα οι ποσοστώσεις δεν θεωρούμε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί το θέμα. Um, Όσον αφορά το θέμα των ε, επιστροφών, τροπολογίες 148-153 γίνεται προσπάθεια να απαλληθεί ο όρος επιστροφής ε, κατά την άποψη της Κομισιόν μια σωστή και καλά εφαρμοσμένη πολιτική επιστροφών ε, ε, είναι ένα από τα μέτρα μέσω των οποίων καταπολεμάται η παράνομη, η παράνομη της καθώς επίσης και η παράνομη μετανάστευση. Στο παράρτημα 2 να υπενθυμίσω ότι αυτές οι δράσεις είναι αυτές οι οποίες έχουν ιδιαίτερα μεγάλη προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία. Οι δύο τροπολογίες επί των ειδικών δράσεων δεν ευθυγραμμίζονται. Είναι η 100 είναι η τροπολογία 184 η τροπολογία 185 η οποία δίνει τη δυνατότητα στις τοπικές αρχές ε, να ε, υποβάλουν έτοιμα χρηματοδότησης ε, για τοπικά μέτρα. Βεβαίως αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε εμάς. Αυτή η ειδική δράση στο παράρτημα 2 αφορά την μοιρασμένη διαχείριση των εθνικών όσον αφορά τα πολιτικών. Όσον αφορά τώρα την ε, κατανομή των κονδυλίων υπάρχουν τροπολογίες 85-86 ε, πρέπει να πω ότι η Κομισιόν έχει εξηγήσει τη μέθοδο υπολογισμού και το ίδιο το αποτέλεσμα των υπολογισμών βρίσκεται στο κείμενο. Έχει ήδη καθοριστεί στο κείμενο λοιπόν προσπαθήσαμε να αποφύγουμε την ε, επιβολή επιπλέον κόστους ε, με τη, μέσω του αιτήματο επιπλέον ε, στοιχείων και υπάρχει όπως είπα και προηγουμένως ένας σαφής τρόπος ο ορισμού. Αυτά ήθελα να σας πω για την ώρα. Για μία ακόμα φορά να σας ευχαριστήσω για την εργασία σας, για την επικοδομητική σας πρόταση κτλ. Ευχαριστώ πολύ. Λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα θα ήθελα να δώσω μια ευκαιρία στο Συμβούλιο, εάν θέλει. ή στους συναδέλφους αν θέλουν να διατυπώσουν κάποια παρατήρηση. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η ομάδα ad hoc εργασίας του Συμβουλίου θα ολοκληρώσει 15 Οκτωβρίου και θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε ε, εντολή από το κορεπέρ του ε, Νοεμβρίου για να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση στο Συμβούλιο σε σχέση με την ε, υπόθεση αυτή επικεντρώνονται στη συζήτηση των εγκάρσεων ζητημάτων που καλύπτουν τις προτάσεις. Το Συμβούλιο συμμερίζεται τη σημασία που αποδίδεται από την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο στα πιο σημαντικά θέματα και η Προεδρία ήδη και θέλουμε να συνεργαστούμε στενά με την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο για να βρούμε λύσεις ταχύτερα δυνατά. Ο στόχος της Προεδρίας είναι η Προεδρία της Κύπρου θα εντείνει τις επαφές για το προσδιορισμό της στρατηγικής, κατά τη διάρκεια της περίοδου των διαπραγματεύσεων και για τον προσδιορισμό της διαδικασίας που θα ακολουθήσουν τα μέρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Παπα-Νικολάου, παρακαλώ, και δεν βλέπω να στείλει κανείς άλλο το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Έχω να αναλάβει την εισήγηση στο θέμα αυτό. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Ευχαριστώ την κυρία Γκυλιόμνα για τη συνεργασία μέχρι τώρα. Την ευχαριστώ. Την κυρία Γκυλιόμ για τη γενικά θετική προσέγγιση. Η θέση μας έτσι προς τους τροπολογίες ότι ενισχύουν και διευκρινίζουν τις διατάξεις. Σε κάποιες αναφορές είμαστε κάπως επικριτικοί, τα έφερε και η κυρία Κιγιόμ, αλλά και η Επιτροπή, πρέπει να τα συστήσουμε και πρέπει να υπογραμμίσω ότι υποστηρίζουμε την κυρία γυγιώμ για το άρθρο 8 ως νομική βάση, με την τροπολογία 17, και θα πρέπει πιστεύω όλες οι πολιτικές ομάδες να συνεργαστούν, να ενωθούν σε αυτό. Άλλα σχόλια. Πρώτον, πρέπει να κοιτάξουμε τι γίνεται με τα κράτη που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. με το ΕΑΖΟ. Να προσφέρουμε ανθρώπινους πόρους και τις προϋποθέσεις του Δουβλίνου. Έχουμε κάνει επίση τροπολογίε και ξέρω ότι είναι ευχερέ. 128, 121, 146 είναι τροπολογίε που αφορούν ειδικέ ιδιαίτερε συνθήκε. Όλοι το γνωρίζουμε τα προβλήματα και θα πρέπει να βρούμε λύσεις με την καταλληλότερη χρηματοδότηση. Θα συζητήσουμε τις συμβαστικές λύσεις και θα καταλήξουμε στεύω σε ένα θετικό αποτέλεσμα εν τέλει. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ την συγκεκριμένη για να Πραγματικά δεν ξέρω αν θα απαντήσω σε όλες τις λεπτομέρειες της Κομισιόν που δεν περίμενα πραγματικά να μπει τόσο πολύ στο ζουμί της ιστορίας. Χρειάζεται να έχουμε ένα ταμείο ισχυρό Όχι μόνο γιατί ε, υπάρχουν ένα σωρό προσδοκίες από το Κοινοβούλιο προς αυτό το σχέδιο, αλλά θα βάλουμε και όλη την ενέργειά μας για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία για το κείμενο. Σας ευχαριστούμε κυρία Γκυγιόμ και τώρα έχει προβλεφθεί στις 26 Νοεμβρίου η συζήτηση στην Επιτροπή μας, ψηφοφορία, είμαστε συμφωνεί, 26 Νοεμβρίου. Και έτσι σε ίσα έχουμε χρόνο να να, βρούμε, να κοιτάξουμε τώρα το σύστημα ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων Eurosur με τον κύριο Μούλντα. και τις σχετικές τροπολογίες. Μόλις 230 τροπολογίες έχουν κατατεθεί στην πρόταση αυτή. Σύντομα κύριε Ντμίλτερ να πάρετε το λόγο γιατί δεν έχουμε πολύ περιθώριο. Έχουμε μόλις μισή ώρα ακόμα για το θέμα σας. Παρακαλώ. Πρόεδρε ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος. Η έκθεσή μου είμαι τυχερός που δέχθηκε θερμή υποδοχή στην ε, Επιτροπή μα. Έχουμε, έχουμε αρκετές τροπολογίες όπως είδατε. πολλέ τροπολογίε με τις οποίες μπορώ να συμφωνήσω. Κύριο στόχος της εκθεσή μου είναι να αποτραπούν τραγωδίες που λαμβάνουν χώρα στη Μεσόγειο. Πολλέ από τι τροπολογίε αφορούν το θέμα αυτό. Κάποιε από αυτέ έχουν βελτιώσει τη θέση μου και θα καλέσω την Επιτροπή να τις εγκρίνει. Και θα επεξεργαστώ συμβαστικές τροπολογίες στο βαθμό του δυνατού. Έτσι ώστε να μην χρειαστεί να ψηφιστούν 280 τροπολογίες χωρίς φορών από την Επιτροπή. Όπως είπα, τις καλωσορίζω τις τροπολογίες στο μεγαλύτερο του βαθμό. Δεύτερο σημείο για την εκθεσία μου χρήση δεδομένων από τη Eurosur με τρίτε χώρε Εγώ επιμένω ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων με τρίτε χώρε. Τα στοιχεία που συλλέγονται θα πρέπει να αναλύονται για να, να χρησιμοποιούνται για να αναλυθεί μια γενική κατάσταση και όχι μια ε, προσωπική κατάσταση να γίνεται προσωποπαγή έρευνα. Τρίτη παρατήρηση, κατάσταση με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Δημοκρατία τη Ιρλανδίας. Έχω, νομίζω, θεωρώ ότι είναι καλύτερο να έχουμε περισσότερες χώρες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό. Υπάρχουν τροπολογίες όπως της Βαρόνης Λάτφορτ, που όμως δεν είμαι βέβαιος εάν μπορώ να τις υποστήριξω, γιατί κάποιες νομικές υπηρεσίες μου είπαν, ή κάποιοι νομικοί εμπειρογνωμόνες μου είπαν ότι υπάρχουν κάποια τεχνικά, νομικά κολλήματα. Εν πάση περιπτώσει θα τα κοιτάξω και θα δω εάν μπορούμε να συμπεριλάβουμε την ε, Βρετανία και την Ιρλανδία στο σύστημα. Με λίγα λόγια, αυτά, κύριε Πρόεδρε, τα περάσματα μου για τις τροπολογίες. Ευχαριστώ κύριε Μίλτερ. Πολύ σύντομα. Η Επιτροπή, δεν βλέπω ποιος κύριος είναι εδώ, σε φάχτ. Ο πρόσωπος Επιτροπής, θέλετε να το λόγο. Ναι, ευχαριστώ. Δύο σύντομες παρατηρήσεις. αφού κοίταξα τις τροπολογίες θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η Eurosur είναι ένα σύστημα που επιδιώκει περισσότερους στόχους, τρεις συγκεκριμένα, την παρεμπόδιση της παράνομης ή της παράτυπης μετανάστευσης, την προστασία των, ε, της ζωής των μεταναστών και των, των, στα εξωτερικά σύνορα και συγκεκριμένα θα ήθελα να αναφέρω τα παραδείγματα στα οποία μπορούμε να εντοπίσουμε αυτού του στόχου. Η Guardia Civil τη Ισπανία αντιμετωπίζει συχνά περιπτώσει ε, μικρών σκαφών που αποπλέουν από τη βόρεια ακτή τη Αφρική και όταν ε, εντοπιστούν, προξενούν ε, ατύχημα, περίπτωση δηλαδή κατά την οποία πρέπει να του παρασχεθεί βοήθεια και έτσι είναι υποχρεωμένε οι αρχέ τη Guardia Civil να προσφέρουν και κατά προτεραιότητα την, ε, τις υπηρεσίες διάσωσης από τους, ε, στους ανθρώπους αυτούς. Ενώ ταυτόχρονα περνούν ε, σκάφη με ναρκωτικά τα οποία δεν είναι σε θέση να συλλάβουν γιατί την ίδια στιγμή είναι υποχρεωμένοι να διασώσουν τους, τους μετανάστες που βρίσκονται στο νερό. Αυτή λοιπόν είναι μια περίπτωση. Μια άλλη περίπτωση οι ζωές των μεταναστών καθίστανται σημαντική προτεραιότητα της Eurosur. Ταυτόχρονα όμως χρειάζονται και τα μέσα που θα μας επιτρέψουν να το υλοποιήσουμε. Και ιδιαίτερα αναφέρομαι στην κοινή υλοποίηση μέσων επιτήρησης όπως δορυφορική επιτήρηση, συστήματα κτλ. Είναι πολλές οι ζωές που θα μπορούσαμε να σώσουμε αν είχαμε την δορυφορική ε, παρακολούθηση και επίσης σε συνεργασία με τις γειτονικέ τρίτες χώρες την πέρα της Μεσογείου θα μπορούσαμε στο πλαίσιο του Eurosur να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα διότι προτείνουμε ακριβώς τα στοιχεία εκείνα που χρειαζόμαστε στην νομοθεσία στον κανονισμό Ευχαριστώ πολύ. Θέλετε το λόγο εκ μέρους της Προεδρίας. Κυρία Γεωργιάδο, έτσι δεν είναι. Ναι, Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγητή και την Επιτροπή. Σημειώνουμε τις θέσεις σας, τις θέσεις που εκφράζετε και τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. και πιστεύουμε ότι θα γίνει ταχύτατα μια ψηφοφορία προς ανατολισμό ώστε να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις πριν από το τέλος της Προεδρίας μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Επίσης, ευπρόσδεκτη την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εγκαθίδρυση του συστήματος και ιδιαίτερα για την για την τήρηση της προθεσμίας της 1ης Οκτωβρίου ως προς την θέση εφαρμογή του συστήματος. Για το ε, έργο για τη δουλειά σε επίπεδο συμβουλίου. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προωθήσουμε το θέμα σε αυτό το στάδιο και έτσι στις προσεχείς εβδομάδες επιδιώκουμε να έχουμε εντολή από το Κορεπέρ ώστε να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσουμε με το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να σας επιβεβαιώσω ότι η Κυπριακή Προεδρία είναι αποφασισμένη να συνεχίσει συνεργασία με τον εισηγητή κύριο τώρα, αλλά και τους σκιώδες, σκιώδες έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια καλή και ισορροπημένη ε, συμφωνία στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ τώρα ποιος θέλει το λόγο, Στούριο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ ήθελα <coughs> να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεσή του με την οποία συμφωνούμε και ελπίζουμε στις επόμενες συνεδριάσεις να ορίσουμε τις ε, λεπτομέρειες ορισμένων ε, πτυχών. Ήδη συναντηθήκαμε, ήταν πολύ ευγενής ο εισηγητής, είχαμε ένα καλό αποτέλεσμα από την πρώτη συνεργασία, οπότε πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε έτσι. Τώρα να υπογραμμίσω κάτι. Μερικά πράγματα ξεφεύγουν από τα πλαίσια της Ευρωσούρ. Όπως ε, ξέρετε, εγώ είμαι Ιταλός και κάθε μέρα, σχεδόν κάθε μέρα έζησα όλα αυτά τα δράματα ε, πνιγμών ε, και ναυαγίων μεταναστών στην Μεσόγειο. Οπότε υπάρχουν μερικές τροπολογίες οι οποίες αναφέρονται στις ε, τροπολογίες υπογραμμίζεται λοιπόν αυτό το, πρόγραμμα, το πρόβλημα. Μετά υπάρχουν και άλλες ε, τροπολογίες ε, οι οποίες στρεβλώνουν την αποστολή της Ευρωσούρα έτσι όπως μας την περιέγραψε και η Κομισιόν με μια τριπλή δηλαδή δράση. Υπάρχουν επίσης και κάποιες τροπολογίες οι οποίες προβλέπουν την εξαφάνιση της παράνομης μετανάστευσης, αλλά αυτό είναι και ο σκοπός ε, της Ευρωσούρ. Μετά υπάρχει και το θέμα των προσωπικών δεδομένων. Και θεωρώ ότι αυτό το οποίο έκανε ο εισηγητής είναι ότι καλύτερο. Διότι υπάρχουν και άλλες τροπολογίες που είναι εκτός θέματος, ίσως η μετάφραση να είναι λάθος. Και αυτός να είναι ο λόγος ίσως που δεν καταλαβαίνω μία τροπολογία που λέει ότι η ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων μέσω του δικτύου ε, της Ευρωσούρ δεν θα πρέπει να αφορούν σε προσωπικά δεδομένα. Πρέπει να είναι αυτό ένα μεταφραστικό λάθος. Δεν μπορούμε να διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα και μετά να μην τα διαβιβάζουμε. Υπάρχει το θέμα το οποίο αφορά στην ε, Μεγάλη Βρετανία και στην Ιρλανδία θα δούμε τι θέση να κρατήσουμε. Αυτό είναι ένα θέμα δηλαδή το οποίο επανέρχεται κάθε φορά που έχουμε ένα μέτρο ε, Σέγγεν ή ένα παρεμφερές μέτρο, όπως είναι η Ιερουσούρ ειναι η ρουσουρ σημερα Θα το ξανασυζητήσουμε όμως και αυτό, είναι ένα λεπτό θέμα το οποίο στο οποίο πρέπει να εμπαθύνουμε καλύτερα. Ευχαριστώ κύριε Σκούρια. Ας προχωρήσουμε στον κύριο Έσιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή γιατί έχει, έχει αναλάβει μια στάση πάρα πολύ επικοδομητική με τους ε, σκεώδεις εισηγητές και αυτό φαίνεται διότι όπως ακούσατε από τους προλαλήσαντες υπάρχει μια απόλυτη συνένεση μεταξύ των πολιτικών ομάδων και της Κομισιόν στο να λεπούνε ότι ένας από τους βασικούς στόχους της Ευρωσούρ θα πρέπει να είναι η διάσωση ανθρωπίν, ανθρώπων. Θα επαναλάβω ίσως αυτό το οποίο είπε ο Ιταλός συνάδελφος. Αυτή η έκθεση πρέπει να είναι συνενετική και όσον αφορά στα προσωπική, στην ανταλλαγή των προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια της Ευρωσούρ. Ο εισηγητής μας παρουσίασε στο, το κείμενό του και εγώ πιστεύω ότι η ανταλλαγή των προσωπικών στοιχείων των πολιτών της Ένωσης θα πρέπει να απαγορεύεται προς τις τρίτες χώρες. Πιστεύω ότι η έκθεση θα είναι εξαιρετική, θα ενισχύσει την Ευρωσούρ και θα βελτιώσει τους στόχους και την αρχιτεκτονική της Ευρωσούρ. Η κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον ε, εισηγητή που έκανε τόσο καλές προτάσεις για τροποποίηση της Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορούμε να δεχτούμε. Έχουμε και μια σειρά τροπολογιών σε τέσσερις τομείς κατά προτεραιότητα τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διάσωση θάλασσα, την προστασία των δεδομένων που παίζουν και τα δύο πολύ σημαντικό ρόλο. Η αδίποτε ανταλλαγή, επεξεργασία ε, δεδομένων θα πρέπει να γίνεται με μια καταχώρηση που θα διατηρεί ίχνη αυτή τη επεξεργασία και ανταλλαγή, ώστε να είναι δυνατόν εκ των υστέρων ακόμη να εντοπιστεί ποιο αντέλαξε με ποιον δεδομένα ή επεξεργάστηκε κατά ποιο τρόπο. Η συνεργασία με τρίτε χώρε. Έχουμε διαγράψει ένα κομμάτι εμεί, διότι θεωρούμε ότι η εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε συνεργασία με τρίτες χώρες δεν γίνεται κατά διαφανή τρόπο. Είχαμε στο παρελθόν ε, τέτοια εμπειρία και προβλήματα στα ανθρώπινα δικαιώματα, παραβιάσεις μάλιστα, με πολλά προβλήματα. Και έτσι δεν θέλουμε να επαναληφθεί αυτό. Γιατί αδίποτε πληροφορία ανταλλάσσεται με τρίτες χώρες μπορεί να οδηγήσει πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα και δεν δεχόμαστε να ε, συμβεί αυτό. Επίσης προτείνουμε διαγραφεί ως προς τα μέσα υποπτίας, γιατί δεν βλέπουμε ουσιαστική απόδειξη ότι χρειάζονται αυτά τα μέσα υποπτίας, που άλλωστε είναι και πολύ δάπανα. Υπάρχει ένας κατάλογος απεριόριστος τεχνολογικών μέσων ε, που ζητούνται και εγώ θα ήμουν μάλλον επιφυλακτική έναντι αυτών των προτάσεων. Η Eurosur είναι ε, εργαλείο, αλλά όχι μόνο εργαλείο για την υλοποίηση άλλων πολιτικών, είναι το ίδιο το Eurosur ε, είδος πολιτικής που κάνει επιλογές για το πώς μπορεί να προστατεύσει τα σύνορά μας, να καταπολεμήσει την παράνομη μετανάστευση, αλλά και άλλες επιλογές και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να μην καταστρέψουμε ή να μην επιτρέψουμε να μεταβληθεί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που όπως είπα είναι και πολύ δάπανη. Επίσης, Frontex. Μιλήσαμε με τον κύριο Λάιτεν σήμερα το πρωί, ο οποίος μας είπε ότι η διάσωση στη θάλασσα είναι για αυτόν κύρια προτεραιότητα. Όταν όμως ρώτησα την Επιτροπή, εάν σκοπεύει να περιλάβει και την διάσωση στη θάλασσα στην ε, εντολή της Frontex, η απάντηση που έλαβα ε, ήταν ότι δεν γίνεται γιατί έσω στη θάλασσα είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ενώ στη Eurosur ρητά αναφέρεται ως προτεραιότητα η διάσωση στη θάλασσα. Πώς κολλάνε όλα αυτά μαζί. Απ' τη μια μας είπατε ότι είναι προτεραιότητα η διάσωση στη θάλασσα, αλλά δεν δίνονται λεπτομέρειες για το πώς θα διασώζονται οι ζωές στη θάλασσα. Άρα λείπει ένα σημαντικό κομμάτι. Και από την άλλη μας λέτε σήμερα το πρωί ότι δεν επιτρέπεται η διάσωση στη θάλασσα ως προτεραιότητα, δεν μπορεί να καταγραφεί ως προτεραιότητα γιατί ανήκει στα κράτη-μέλη και όχι στην Επιτροπή. Επομένως όλα αυτά πώς θα εξηγηθούν. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσω την απάντηση. Γιατί είτε έχουμε διάσωση στη θάλασσα ως προτεραιότητα, χωρίς κανένα νόημα και παραμένει στο προήμιο, είτε υπάρχει ουσιαστική αρμοδιότητα και τότε πρέπει να ξεχωρίσουμε την κατάσταση σχέση με τα κράτη-μέλη. Πάντως είναι όλα πολύ συγκεκριμένα. Ευχαριστώ. κύριος παρακαλώ. Δεν είχατε στήσει το λόγο. Καλά. Κύριε Ένστ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Μια πολύ δύσκολη έκθεση και πτυχές που έχει εξετάσεις που μας φέρονται τόσο σημαντικές. Είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρχει ανταλλαγή απόψεων με τα τρίτα κράτη. Και γενικά η διάσωση είναι μια πολύ καλή ιδέα, αλλά μέχρι εκεί, μέχρι εκεί πάει η θετική μας αποτίμηση. Της εκθέσεως ουσιαστικά, ε, γιατί το Eurosur για μας είναι αμφισβητήσιμης αξίας. Το λέω ομά. Το απορρίπτουμε για διάφορους λόγους. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι σήμερα το πρωί ακούσαμε έναν συνάδελφο από τη Frontex που μας είπε διάφορα πράγματα για την διάσωση και το τι μπορούν να κάνουν ακόμη για τη διάσωση, για το τι διπράττουν κτλ. Αλλά τότε δεν χρειάζεται αυτό το σύστημα αποπτίας, χρειάζεται ένα σύστημα διάσωσης αλλά όχι επιτήρησης με τον τρόπο αυτόν που διαμορφώνεται και περιγράφεται στο άρθρο 12. Επίσης, το πρόβλημά μας, για να πούμε στις λεπτομέρειες, δεν είναι η καταπολέμηση της περσινοριακής εγκληματικότητας, αλλά το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης. Έχουμε ακούσει διάφορους όρους εδώ, παράτυπη, παράνομη, μιλάθρο μετανάστευση. Κανένας από αυτούς δεν είναι ικανοποιητικό. Εδώ λοιπόν η, η έννοια, αλλά πάνω απ' όλα για λόγους ουσίας και περιεχομένου, είναι για μας απορριπταία της παράνομης μετανάστευσης. Επίσης, Πουθενά δεν αναφέρεται ότι δεν αναφέρονται λόγοι και αποδείξεις γιατί χρειάζεται ένα τέτοιο σύστημα. Φερρυπίν. Τα μη επανδρομένα αεροπλάνα, τα drones. Γιατί τα χρειαζόμαστε για να εντοπίζουμε τέτοιου είδους ε, κινήσεις ε, ενδεχομένως παράνομων μεταναστών. Εγώ νομίζω ότι εδώ πρόκειται απλώς για μια προσπάθεια των λόμπι, ένα πρόγραμμα των λόμπι και γι' αυτό και απορρίπτουμε ρητά τις θέσεις αυτές. Θα δείτε ότι έχουμε κάνει και μια τροπολογία όπου ρητά λέμε ότι απορρίπτουμε την πρόταση. Ξέρουμε βεβαίως ότι θα δημορφωθούν διαφορετικά οι πλειονότητες, ωστόσο παραμένουμε στη συζήτηση. για να επιδιώξουμε να βρούμε κάποιες λογικές και συνεπείς με το στόχο της διάσωσης των ζώων μεταναστών λύσεις. Αλλά δεν θέλουμε ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων με τον τρόπο που παρουσιάζεται εδώ. Αυτά τα συστήματα επιτήρησης και σημειώνω ότι ε, κομμάτια μόνο του άρθρου 12 έχουμε απαλείψει από το κείμενο και δεν έχουμε προτείνει τη διαγραφή ολόκληρου του άρθρου. Ε, πρέπει λοιπόν να απευθύνονται αυτές οι προσπάθειες όλες στον στόχο της διάσωσης στη θάλασσα ιδιαίτερος και θα προσπαθήσουμε στο βαθμό του δυνατού να συνεργαστούμε σε συμβουλευτικές τροπολογίες. Αυτά κατά τα άλλα για την ε, τεχνολογία της επιτήρησης. Αν σκεφτούμε ότι υπάρχουν τα εθνικά μέσα και το, τα ευρωπαϊκά μέσα. Πάντα υπάρχουν δυνατότητες επιτήρησης χωρίς να χρειάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιτήρηση. Εδώ και το λέω χωρίς να έχει ιδιαίτερη σημασία ίσως, αλλά υπάρχει ένας κίνδυνος εκτεταμένης ε, παρακολούθησης και γι' αυτό και απορρίπτουμε το κείμενο το συγκεκριμένο, ιδιαίτερα γιατί τη διατύπωση του φαίνεται πολύ ύποπτη. Ευχαριστώ. Κύριε Ένστα, θα ξανακούσω την Επιτροπή πριν περάσουμε στον εισηγητή για να καταλήξουμε. Ήθιστε η Επιτροπή να σχολιάζει τα, τις παρατηρήσεις. Ο εκπρόσωπος Επιτροπής, κύριο Ζήφαρτ, παρακαλώ. Thank Ευχαριστώ. Νομίζω ότι απλώς θα επαναλάβω αυτά που είπα και προηγουμένως. Η προστασία της ζωής των μεταναστών είναι σοφής μας στόχος. Πρέπει να σταματήσει πια ε, αυτή η ιστορία με τους ε, μετανάστες που πνίγονται και χάνουν τη ζωή τους στη Μεσόγειο. Από την άλλη πλευρά η ε, έρευνα και η διάσωση δεν είναι θέμα αρμοδιότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως υπάρχει συνεργασία με την διεθνή ε, θαλάσσια ε, με τον Διεθνή Οργανισμό IMO και βεβαίως υπάρχει και η κοινή ε, οργάνωση της αντιμετώπισης ε, των ατυχημάτων ή των ε, καταστάσεων κινδύνου στην θάλασσα αλλά μπορεί να είναι και ατύχημα ενός κουρασγερόπλιου ή μπορεί να είναι το ναυάγιο ενός πετρελαιοφόρου κτλ. Ε, πρέπει οι αγωνομικής απόψεως να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Γι' αυτό λοιπόν έχει διατυπωθεί η πρόταση ως ε, ε, την έχετε μπροστά σας και όπως την έχετε μελετήσει. Όσον αφορά το θέμα των μικρών σκαφών σε σχέση και με το άρθρο 12. Η Eurosur δεν είναι επενδυτικό πρόγραμμα για τη βιομηχανία, όμως στοχεύει στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας ε, κάθε μορφής ε, ε, επιτήρησης σε συνεργασία με όλα τα όργανα. 20 άρθρα ασχολούνται με την διοργανική συμφωνία, συνεργασία, συγγνώμη, τη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών. Ένα άρθρο ασχολείται με το άρθρο 12, με την τεχνολογία ε, της ε, επιτήρησης Ε, και υπάρχει ειδικό ε, εξοπλισμός όσον αφορά την ανείχνευση ε, των μικρών και διάσωση των μικρών σκαφών που κυρίως αυτές, αυτά τα μικρά σκάφη ευθύνονται για τον πνιγμό των ε, παρανόμων μεταναστών. Υπάρχουν επίσης και ελικόπτερα και άλλα ε, σκάφη περιπολίας ε, και βεβαίως εμείς θέλουμε από μια διαδικασία που απαιτεί πολλά, πολύ μεγάλο εξοπλισμό και πολλά μέσα θέλουμε να περάσουμε σε ένα άλλο σύστημα πιο ευφιές το οποίο θα μπορεί να βρει τα μικρά αυτά σκάφη και πιστεύουμε ότι η κοινή εφαρμογή των εργαλείων επιτήρησης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ωστόσο, ε, γίνεται πάντα λόγος ε, σε αυτά τα ε, μη επανδρομένα αεροσκάφη τα οποία όμως δεν μπορούν να κάνουν πτήσεις πάνω από αστικές περιοχές. Παίρνει πολύ χρόνο η ενεργοποίησή τους και επομένως ε, απλώς αναφέρθηκε με την έννοια ότι δεν θέλουμε να το αποκλείσουμε για τα επόμενα πέντε χρόνια αλλά δεν είναι η κύρια επιλογή για τα επόμενα ε, χρόνια και οπωσδήποτε ε, σας λέω η χρήση είναι δύσκολη η χρήση που γίνεται για αυτόν τον μη επανδρομένων πτήσεων σε άλλα μέρη του κόσμου έχει τελείως διαφορετικό σκοπό και δεν μας καλύπτει. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Μούλτερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Σκουρία ότι ο στόχος της πρότασης δεν είναι μονάχα να σώσει ανθρώπινες ζωές, αλλά ε, αυτό βεβαίως το στοιχείο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Αλλά υπάρχει και άλλο περιεχόμενο, δεν το λησμονούμε. Κυρία Καρα, μπορώ να σας πω ότι όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, ε, ένας από τους κύριους στόχους μου είναι να μην υπάρχει δυνατότητα συλλογής ε, δεδομένων. Αυτό είναι ένα ασθενέ σημείο του συστήματος. Θα πρέπει να γίνεται ε, ερμηνεία των μαζικών δεδομένων και όχι ανάλυση ατομικών προσωπικών δεδομένων. Όσον αφορά την επιτήρηση, θα δω το κεφάλαιο αυτό. Σε γενικές γραμμές πάντως μπορώ να πω ότι και άκουσα και σήμερα το πρωί τον ε, διευθυντή της Frontex το κύριο πρόβλημα είναι τι συμβαίνει από τη στιγμή που έχετε ανακαλύψει, έχετε βρει, έχετε εντοπίσει ένα μικρό σκάφος ε, με πολλούς ε, παράνομους μετανάστες. Τι γίνεται τότε. Ε, δεν μπορεί αυτός ο κόσμος να είναι αρμοδιότητα της Eurosur. Θα, θα είναι αρμοδιότητα του κράτους μέλους. Θα τα διαβάσω όλα αυτά, θα τα ξανακοιτάξω. Εγώ επανειλημμένα έθεσα το σχετικό ερώτημα στον ε, ε, διευθυντή της Frontex σήμερα το πρωί, αλλά δεν είχα έτσι και πολύ καλή απάντηση. Πάντως, να σας πω ότι θα υποβάλω τη συμβαστική μου πρόταση και εν πάση περιπτώσει την τελική κρίση θα την αναλάβει ε, μέσω ψηφοφορίας η Επιτροπής μας. Πάρα πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε για την εργασία που κάνατε, για τη θέση που πήρατε για μία ακόμα φορά. Δεν ξεπεράσατε το χρόνο σας, είσαστε, είσαστε ακριβείς, είσαστε ε, σύντομος. Ψήφος προσανατολισμού 26-27 Νοεμβρίου. στην επόμενη τακτική μας συνεδρίαση τον Νοέμβριο. Πολύ ωραία. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο που αφορά το ε, Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Ο κύριος Λορέντσο Φοντάνα είναι εισηγητής. Όμως στην πρόταση αυτή περιέχει διατάξεις οι οποίες ε, θα, αρχίσουν, θα αρχίσουν να ισχύουν, να ισχύουν από το 14 ε, μέχρι 16. Πολλές είναι οι τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. Θα δώσουμε το λόγο αμέσως στον εισηγητή και μετά Κομισιόν και Συμβούλιο. Κύριε Φοντάνα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για το ενδιαφέρον τους και όπως ανήγγειλε και ο πρόεδρος έχουν παρουσιακατατεθεί πολλές τροπολογίες. Και φυσικά εγώ μαζί με τους και όλες οι συγητές, θα, θα κοιτάξω να περάσω τις περισσότερες, κυρίως αυτές που τίνουν προς την απλούστευση και τη διαφάνεια στη χρήση των κονδυλίων και στη βελτίωση της διαδικασίας ενημέρωσης. Εμείς προσπαθήσαμε σε αυτήν την ε, προσπαθήσαμε σε αυτήν την έκθεση να εξάρουμε το ρόλο που θα μπορούσαν να παίξει η τοπική αυτοδιοίκηση ώστε να τονιστεί η αρχή της ε, επικουρικότητες και σε αυτό το πλαίσιο. Και, θεω... και ξέρουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές ένομες τάξεις ανά την Ευρώπη. Αλλά αυτό θα, το σημείο είναι πολύ σημαντικό. Αν χρησιμοποιηθεί ως ένα μέσο το οποίο δεν θα γραφειοκρατικοποιήσει παραπάνω αλλά θα πλουστεύσει τη διαδικασία. Εμείς συναντηθήκαμε με, το, με τους υπαλλήλους και με τους και όδης και τους ευχαριστώ. Υπάρχουν ορισμένα σημεία για τη γύρω από τα οποία θα πρέπει να βρούμε μία λύση. Ε, τροπολογίες της κυρίας Κέλλερ ε, που θέλει να καταργήσουμε τις δράσεις σε τρίτες χώρες που θα είναι χρηματοδοτημένες από τις, ε, ε, από τις εσωτερικές υποθέσεις. Τώρα έχουμε ένα ζήτημα με την τροπολογία 69. όταν ε, ζητεί το να δημιουργηθεί μία ομάδα εργασίας η οποία, την οποία θα πρέπει να συμβουλευόμαστε για δράση σε τρίτες χώρες. Αυτή η τροπολογία έχει θετικές πλευρές στο βαθμό που θα μπορούσαμε να εμπλέξουμε σε αυτή την ομάδα εργασίας και την κοινωνία των πολιτών και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Θα πρέπει όμως να προσέξουμε ώστε αυτό να μην καταστεί ένα, ένα πρόβλημα καθυστερήσεων και κολλησιεργιών για τις τρίτες χώρες. Και γι' αυτό Θέλαμε να ρωτήσουμε και την Κομισιόν η οποία μας είπε ήδη δηλαδή ότι κάτι τέτοιο ήδη υφίσταται αλλά να μας δώσει παραπάνω διευκρινήσεις. Ένα άλλο σημείο για το οποίο θα πρέπει να βρούμε έναν συμβιβασμό είναι το θέμα της συγχρηματοδότησης. έχουμε διάφορες τροπολογίες σχετικά. Άλλοι λένε 75%, άλλοι 80%, άλλοι 100% και συγχρηματοδότηση και η Κομισιόν λέει επίσης 100% συγχρηματοδότηση. Πρέπει να βρούμε μια συμφωνία όμως να δούμε ποια είναι η καλύτερη θέση. Γιατί καλό είναι τα κράτη-μέλη να έχουν ευθύνες αλλά δεν πρέπει και πριν ορίσουμε τα ποσοστά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τι γίνεται σε περίπτωση που έχουμε ένα κατεπήγον. Τώρα, θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία στις διάφορες ευαισθησίες που προέκυψαν από τη συνεδρίαση των σχεδόν εισηγητών. Τώρα ένα σημείο που δημιούργησε κάποιο πρόβλημα είναι οι τροπολογίες 127 και 72. Μεταξύ των άλλων Ζητήσαμε και την ε, νομική, ε, προσφύγαμε μάλλον στην νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου για να μας συμβουλεύσει διότι ορισμένες ε, εκτελεστικές πράξεις μετατρέπονται σε κατεξουσιοδότηση πράξη. Στην 127 τροπολογία καταλάβαμε και από την νομική υπηρεσία επίση, το καταλάβαμε, ε, ότι όσα γράφει η Κομισιόν είναι νομικός ορθά, αλλά για την 72 έχω κάποιο πρόβλημα. Διότι η πρόταση της Επιτροπής αφήνει ορισμένες αμφιβολίες, διότι ε, ναι εντάξει εμείς ε, πρέπει να σεβόμαστε το άρθρο 290 της συνθήκης, αλλά όμως θα πρέπει να δούμε πώς η διακριτική ευχέρεια αφήνουμε στην Κομισιόν. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό με τον καλύτερο τρόπο. Φυσικά οι τροπολογίες είναι πολλές, αλλά με καλό πνεύμα συνεργασίας όλων των σκιωδών εισηγητών, θα προχωρήσουμε, θα έχουμε και άλλες συνεδριάσεις και θα δούμε ποια τελική μορφή θα πάρει αυτή η έκθεση. Ευχαριστώ κύριε Φοντάνα. Τώρα η Κομισιόν και η Προεδρία. Η κυρία Μπελίντα Πάικ από την Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τον εισηγητή θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, ε, Επιτροπή για αυτόν τον κανονισμό που όπως είπα και προηγουμένως συνδυάζεται με το Ταμείο συνδυάζει με το Ταμείο την Άσυλο και τη Μετανάστευση με το Ταμείο για την Εσωτερική Ασφάλεια. Έχουμε κάνει γενικές προτάσεις τις οποίες έχουμε εξηγήσει και σε προηγούμενη συνάντηση με την οποία όταν συζητήθηκε ο κανονισμός. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ε, απλούστευση και νομίζω ότι η απουσία τροπολογιών σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει ότι έγινε μια προσπάθεια. Ε, βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει και κάποια προσαρμογή σε σχέση με τον χρηματοδομητικό κανονισμό. Πρώτα απ' όλα να αναφερθώ σε ορισμένα από τα σημεία τα οποία έθιξε ο ίδιος ο εισηγητής για την εξωτερική διάσταση υπάρχουν δύο σημεία. Ένα, ότι πρέπει να υπάρχει εξωτερική διάσταση και δεύτερο σημείο, πώς μπορούμε να αποκαταστήσουμε την συνοχή με εξωτερικά, με την εξωτερική διάσταση. Νομίζω ότι ο εισηγητή μου ζήτησε να εξηγήσω γιατί πρέπει να υπάρχει εξωτερική διάσταση. Θα, μπορούσαμε να, θα μπορούσα να μιλάω ώρες για αυτό το θέμα αλλά νομίζω ότι ε, υπάρχουν οι φύση τα δελτία και η φύση, ε, το δελτίο 13 ασχολείται με το θέμα αυτό και είναι ε, καθιστά πάρα πολύ σαφές τον λόγο, σαφή συγγνώμη, τον λόγο για τον οποίο υπάρχει εξωτερική διάσταση και στην ίδια φύση, στο ίδιο δελτίο δίνουμε παραδείγματα για τις δράσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν δράσεις οι οποίες αποβαίνουν προς όφελος όλων των πολιτών κρατών της Ευρώπης και εντάσσονται στην εσωτερική και όχι την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε να επανέλθουμε βεβαίω στο θέμα της εξωτερικής δράσης, αλλά παραμένει ε, πεποίθησή μας ότι ε, έπρεπε υπό το νέο ταμείο, κυρίως όσον αφορά την άμεση χρηματοδότηση, θα έπρεπε να είμαστε σε θέση να χρηματοδοτήσουμε δράσεις και σε σχέση με τι τρίτε χώρε, γιατί αυτό ήταν κάτι που έλειπε από τον προηγούμενο ε, κανονισμό. Ο συντονισμό επίση, ε, πώ επιτυγχάνουμε συνοχή με άλλες εξωτερικές πολιτικές, ε, πώ μπορούμε να επιτύχουμε καλύτερο συντονισμό. Οφείλω να πω ότι δεν συμφωνούμε με τις τροπολογίες οι οποίες ε, είναι πολύ αναλυτικές και αναφέρονται σε κάθε λεπτομέρεια ε, στο τι πρέπει να κάνει η Κομισιόν και τι πρέπει να προβλέψει η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Υπάρχουν μηχανισμοί εσωτερικού συντονισμού και όχι μονάχα για τις εξωτερικές δράσεις. Ε, θα πρέπει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής να είμαστε σίγουροι ότι και για το, για το άσυλο και την μετανάστευση, ε, όλες ε, οι δράσεις ε, είναι συνεκτικές, ας πούμε, με το κοινωνικό ταμείο. έχουμε τρόπους και τους αναφέρουμε για τον τρόπο με τον οποίο θα οργανωθούν οι υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τροπολογία 36 και τροπολογία 9 από την Επιτροπή Προϋπολογισμών ασχολούνται με τις αιτιολογικές σκέψεις προτείνω ότι ενδεχομένως ε, ότι θα μπορούσε να γίνει μία προσθήκη στην αιτιολογική σκέψη 6 και να λέει για να διασφαλιστεί αυτή η συνοχή, κόμμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με την ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης θα χρησιμοποιήσει πλήρως τους ισχύοντες μηχανισμούς και θα τους ενισχύσει εάν και όπου δει. Βεβαίω θα στείλω το κείμενο αυτό στον εισηγητή, να δούμε αν τον βοηθάει, αλλά νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό μπορούμε να ανταποκριθούμε σε ορισμένα αιτήματα, σε αριθμό ε, ε, ε, αιτημάτων τα οποία περιλαμβάνονται και σε τροπολογίε. Νομίζω ότι καλύτερα να κάνουμε την τροποποίηση στην αιτιολογική σκέψη, όχι στα άρθρα. Επίσης υπάρχουν και άλλες τροπολογίες οι οποίες αφορούν με την υλοποίηση από δράση της Επιτροπής, κυρίως τροπολογίες 72, 107 και 131. Η Κομισιόν δεν μπορεί να δεχτεί τις τροπολογίες αυτές. Η αλλαγή, η αντικατάσταση μάλλον των εκτελεστικών πράξεων από κατεξα από κατεξουσιοδότηση πράξης ε, θα μπορούσε να δημιουργήσει ε, προβλήματα και τα οποία θα φανούν οπωσδήποτε στην ε, ενδιάμεση αναθεώρηση. Νομίζω ότι οι εκτελεστικές πράξεις είναι το σωστό εργαλείο και φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσει και το Συμβούλιο. Η Κομισιόν επίσης αποφάσισε να ακολουθήσει στενά την ε, κοινή κατανόηση των ε, θεσμικών οργάνων. Και θα δούμε βεβαίως εάν ε, θα προκύψει κάποια αποκλίνουσα άποψη και η νομική υπηρεσία σε αυτή την περίπτωση θα είναι σε θέση να μας εξηγήσει. 72, 107, 131 τροπολογίες δεν γίνονται δεχτές. Να πω και μερικά άλλα σημεία, αν μου επιτρέπετε. Εταιρική σχέση. Καλωσορίζουμε το ενδιαφέρον που δείχνεται για αυτήν. Πιστεύουμε ότι ε, είναι πολλοί αυτοί που πιστεύουν ότι πρέπει να είναι καλύτερα δομημένη η εταιρική σχέση, αλλά θα πρέπει να ε, παραμείνει σε ένα ε, λογικό μέγεθος έτσι ώστε να είναι διαχειρίσιμο. Βεβαίως, οι υπηρεσίες, ε, ε, οι διάφορες υπηρεσίες οπωσδήποτε θα εμπλακούν στις διαδικασίες. Οι τροπολογίες οι οποίες ε, αντιμετωπίζουν το θέμα του, της ροής του, του ρευστού σε την, από τα κράτη-μέλη ε, και η κοινή διαχείριση του ε, Ταμείου καθώς επίσης ε, και οι πληρωμές. Αυτά όλα είναι σημεία τα οποία θα συζητηθούν σε υψηλότερο επίπεδο, αλλά βεβαίως θα συζητηθούν και στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου. Όσον αφορά το άρθρο 5, υπάρχουν εκεί διάφορες τροπολογίες οι οποίες έχουν υποβληθεί. το πολιετές πλαίσιο, όχι μονάχα σε αυτό το σημείο αλλά και σε άλλα, μας υποχρεώνει να παραμείνουμε σε συγκεκριμένες ε, γραμμές. Τέλος, ε, υπάρχει τροπολογία 113 πρόταση να δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, το, προ, το προσχέδιο του προγράμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν αντιτίθεμαι σε αυτό. αλλά ίσως πιο καλό θα ήταν ε, από το, για το Κοινοβούλιο να πάρει αντίγραφα των εγκεκριμένων προγραμμάτων. Βεβαίως ε, θα σας δώσω κύριε Ισηγητά και τις ε, προτάσεις Κιμάνου που έκανε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η Προεδρία παρακαλώ θέλει να κάνει μια παρέμβαση. Έχετε το λόγο. Όπως είπα και νωρίτερα στην παρέμβασή μου για την πρόταση για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, η ομάδα ad του Συμβουλίου θα ολοκληρώσει την ε, πρώτη φάση στις 15 Οκτωβρίου. Και έτσι αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο επικεντρώνεται στις συζητήσεις όλων των εγκάρσιων θεμάτων που διέπουν τις ε, τέσσερις προτάσεις κανονισμού, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, η Προεδρία ήδη έχει ευθυγραμμίσει την ε, συμβαστική της πρόσταση στα σχετικά αρθρά του, των προτιμωμένων κανονισμών με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Ιδιαίτερα οι προτάσεις παρατηρήσεις Επιτροπής και του Κοινοβουλίου για ασθενή συνεργασία με Επιτροπή και Κοινοβούλιο κατά τις επίσημες διαπραγματεύσεις για τον τριμερι, του τριμερούς διαλόγου θα μας οδηγήσουν πιστεύουμε σε ένα καλό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου στον τομέα της, ε, των εσωτερικών. Και της μετανάστευσης ευχαριστώ πολύ. Κύριος Φως. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εκ μέρους του κ. Πέρκαρ, του σκιώδου συγητού που δεν μπορούσε να έρθει σήμερα. Θα ήθελα εκ μέρους της πολιτικής μου ομάδας να τοποθετηθώ στο άρθρα 3 και 14, εκεί όπου γίνεται λόγος για την προσθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα τις τροπολογίες της κυρίας Φαζόν και της Φρανσίσκα Κέλλας Με την προστιθέμενη αξία και την επαλήθευσή της στα εθνικά προγράμματα. Διότι θεωρούμε ότι η τροπολογία 55 της κ. Φαζόν είναι μια καλή περιγραφή για την ε, προστιθέμενη αξία και έτσι πιστεύουμε ότι μπορούμε να βρούμε μια συμβαστική λύση στα άρθρα 5 και 25 ε, απρόβλεπτη, απροειδοποίητη έλεγχη κ. Σπίρκερ αλλά και οι άλλοι έχουν κάνει τροπολογία, τροπολογίες που τροποποιούν κάπως την πρόταση αυτή των ε, ε, απρόβλεπτων των μη ανακοινωθέντων ελέγχων, που είναι μια έννοια ουσιοδέστατη σημασία για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, και όμως ε, δεν φαίνεται πάντοτε τόσο αυτονόητο να υλοποιηθούν γιατί ε, διατυπώνουμε συνήθως στο κείμενο την ιδέα του where appropriate, όπου δει, όπου χρειάζεται, όπου είναι σκόπιμο ως προϋπόθεση για να διεξαχθούν αυτοί οι έλεγχοι. Για το 6α και τη χρηματοδότηση σε σχέση με τρίτα κράτη έχουμε περισσότερες δυσκολίες δεν βλέπουμε τρόπο, δεν υπάρχει βάση για να συμφωνήσουμε πάνω στο άρθρο αυτό. Η 69 τροπολογία των Σοσιαλιστών Δημοκρατών προβλέπει μέτρα σε σχέση με τρίτα κράτη και συνεχίζει για να φτάσει μέχρι την ενοποίηση. Πράγμα το οποίο μας, μας ε, προξενεί αρκετές δυσκολίες και δισταγμούς, όσο προς το τι μπορεί να σημαίνει αυτό αλλά και η εσωτερική οργάνωση, οι δομές της Επιτροπής κτλ. δεν θα πρέπει, πιστεύουμε, να, διέπονται, να ρυθμίζονται μέσα από έναν κανονισμό. Μια ομάδα εργασίας μπορεί να προσφέρει κάτι ουσιαστικό. Ε, εμείς μόνο προτάσεις θεωρούμε ότι μπορεί να διατυπώνει, αλλά όχι με υπερβολικό γραφειοκρατικό φόρτο. Τέτοιες δομές ωστόσο δεν ξέρουμε αν υπάρχουν, αν μπορούν να προβληθούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για την άμεση βοήθεια, άρθρο 8, υπάρχουν πάλι προτάσεις σε σχέση με το ύψος της άμεσης βοήθεια 100%. 80%, 90%, 75%. Εδώ νομίζω ότι με όλες τις προτάσεις που κατευθεί μπορούμε να βρούμε μια καλή συμβαστική λύση για το άρθρο 12 την εταιρική σχέση, αλλά και τον πολιτικό διάλογο. Παρακάτω, ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε στο να διαφυλαχτεί, να διατηρηθεί η δομή που σκοπεύει να θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρθρο 12. Φάση της ανάπτυξης και της υλοποίησης των εθνικών προγραμμάτων. Είμαστε εταίροι όπως και οι περιφερειακές αρχές και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις για το Συμβούλιο για να γνωμοδοτούμε, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια ευελιξία ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ανησυχίες και τα μέληματα των κρατών μελών. πολιτικός διάλογος μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 100 μελών. Για λόγους ε, πρακτικής εφαρμογής πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερως ώστε να μην εισαγάγουμε και άλλους φορείς ε, και δομές είτε ιδιωτικού είτε δημόσιου χαρακτήρα. Άρθρο 16, παράγραφος 5 τροπολογία σε σχέση με, ε, με πρόταση διαγραφής του άρθρου αυτού του κ. Κίρκοπ με δυνατότητα αύξηση του ποσού στο 90%. Εμάς, ως ΕΛΚ, μας φαίνεται μάλλον αντιπαραγωγική αυτή η πρόταση. αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στο σχετικό προπολογισμό της Ένωσης. Οι αιτιολογημένες ε, προϋποθέσεις ή όροι νομίζω πρέπει να εξεταστούν. Μετά στο άρθρο 3, προχρηματοδότηση όπου προτείνεται ετήσια προχρηματοδότηση ύψους 2,5% του συνολικού ποσού ενός εθνικού προγράμματος. που πολλά κράτη-μέλη θεωρούν πως δεν είναι πλέον υλοποιήσιμο. Είναι πολύ ψηλό το ποσό. 51, άρθρο 51 δημοσιοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης, όπου και πάλι μπορεί να βρεθεί συμβαστική λύση. Σημαντικό είναι εδώ να μην προκύπτει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, για την ε, κρατική ασφάλεια και τη δημόσια τάξη. Ίσως λοιπόν μια διάθεση αυτοπεριορισμού μπορούμε να βρούμε συμβαστικές λύσεις και επίσης η 73 και 127 των σοσιαλιστών δημοκρατών της κυρίας Φαζόν. Εδώ, εάν ζητήσουμε γνωμοδότηση από νομική υπηρεσία, θα πρέπει αντίστοιχα να καλύψει και τους άλλους κανονισμούς για να έχουμε μια γενική θεώρηση και να είμαστε θέσεις να τα αξιολογήσουμε όλα. Κυρία Φαζόν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Εγώ πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Φοντάνα για την δουλειά του και την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Τώρα, στην πολιτική μας ομάδα εμείς θέλαμε να βελτιώσουμε κυρίως την διαφάνεια και θέλουμε σε αυτήν την πρόταση να συμπεριλάβουμε όσο των δυνατόν περισσότερους πρωταγωνιστές, κοινωνία των πολιτών, κοινοβούλιο κλπ. κλπ. Από αυτά που ακούσαμε σήμερα, το πιο καυτό σημείο είναι αυτό της χρηματοδότησης στις τρίτες χώρες. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε συγκεκριμένα κανάλια χρηματοδότησης για τη χρηματοδότηση αυτών των δράσεων, και οι τροπολογίες της ομάδας μας τίνουν προς την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής της Κομισιόν μάλλον για να, και να μπορέσουμε να εγγυθούμε και ένα συντονισμό από την ε, από, τον οργαν... από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Θεωρούμε θεωρούμε ότι δεν χρειάζονται παραπάνω δαπάνες. Πρέπει να έχουμε ένα συντονιστικό όργανο το οποίο θα συντονίζει τις δράσεις στις τρίτες χώρες. Ακούσαμε ότι η Κομισιόν έχει ένα μηχανισμό αυτού του τύπου στη διάθεσή της. Εγώ όμως δεν το βρήκα στην ε, έκθεση. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ζητήσουμε εγγύσεις όσον αφορά το 72 και το 127 για τις κατεξουσιοδότης πράξεις, τόσο για το πρόγραμμα εργασίας όσο και για τα εθνικά προγράμματα, θα ήθελα να ζητήσω μία επίσημη γνώμη της νομικής υπηρεσίας. Εμείς χρειαζόμαστε μια, κοινή, μια συνολική και μια σφαιρική μάλλον επίσημη γνώμη. Τώρα εμείς ακούσαμε χθες ότι αυτή η έκθεση συντάχθηκε πολύ διαστικά, οπότε πρέπει να την συζητήσουμε. Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη θα πρέπει να έχουν και μια λύση και μια αξία, αλλά κυρίως να έχουν μια ευκταία λύση για την προστιθέμενη αξία. Θα πρέπει να πετύχουμε αυτά αποτελέσματα για την ασφάλεια και από τη χρήση αυτών των κονδυλίων, για τη συγχρηματοδότηση. Θεωρούμε ότι η συγχρηματοδότηση σε ειδικέ περιπτώσεις αλλά και συγκυριακές, ε, δικαιολογημένες συγκυριακές περιπτώσεις, η χρηματοδότηση πρέπει να προσεγγίζει το 90%. Όταν έχουμε δηλαδή πολύ σοβαρές καταστάσεις θα πρέπει να προβλέπουμε τη χρηματοδότηση 100%. Κυρίως άμα δούμε την ε, χάλια οικονομική κατάσταση σε ορισμένα κράτη της Ένωσης. Εμείς ε, δεν θα πρέπει να καταλήξουμε σε μία κατάσταση όπου δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε και τα θύματα είναι οι πολίτες οι ίδιοι. Εγώ τρέφω εμπιστοσύνη ότι θα έχουμε μια επικοδομητική συζήτηση για αυτά τα σημεία και θα βρούμε μια ευφύ Κυρία Κέλλερ. Και μετά η συγκεκριτρία. Ευχαριστώ. Μετά η συγκεντρία. Δεν θέλω να επανέλθω στα όσα είπα πριν και χτες. Για τον προϋπολογισμό ήδη αναφέρθηκε. Για τις τρίτες χώρες δεν ε, θέλουμε να πούμε ότι είμαστε κατά των τρίτων χωρών, αλλά απλώς αυτή η πίστοση για πρώτη φορά εμφανίζεται στον προϋπολογισμό των εσωτερικών και πρέπει με πολύ μεγάλη σύνεση να τη χειριστούμε. πολλά θέματα σχετικά με τις χώρες ήδη μπορούμε να τα πράξουμε, αλλά υπαγόντας την υπηρεσία εξωτερικής δράση ή τη Γενική Διεύθυνση για την Ανάπτυξη. Δεν μπορεί κανείς δηλαδή να συνδυάσει μετανάστευση με δράσεις. Υπάρχουν ε, οι αιτούντες στο άσυλο και όλο το σύστημα οικοδόμησης ε, ε, συστημάτων υποδοχής και όλα αυτά δεν χρειάζεται λοιπόν να τα αναφέρουμε αυτά για να μην μπερδέψουμε περισσότερο το κείμενο. Έστω και αν θέλει η Επιτροπή κάποια πράγματα να τα ξεκαθαρίσει. Δεν είμαστε λοιπόν υπέρ αυτή τη ε, ειδική του στον προπολογισμό. Να μην φαίνεται δηλαδή ότι αυτομάτω δεν τίθεται τα ποσά αυτά. Και κατόπιν πολύ ορίμου σκέψεως καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι δεν θέλουμε αυτές τις λύσεις. Ελπίζουμε να μας ακολουθήσετε. Θέματα σημαντικά για μας ε, είναι η διαφάνεια που ανέφεραν αρκετοί και ίσως μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει αν υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με τα όσα είπε ο κύριος Φως για θέματα ασφάλειας που εμείς θεωρούσαμε ότι καλύπτονται από τους γενικούς κανόνες περιεγράφων εκτό εκτός και αν μας πει η Επιτροπή κάτι διαφορετικό για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις και ιδιαίτερα την τροπολογία 72 που έχει μεγάλη σημασία. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα είναι να προσδιορίσουμε δείκτες για τα εθνικά προγράμματα. Και εδώ λοιπόν ζητείτε σαφήνεια στους δείκτες. Ομάδα εργασία των σοσιαλδημοκρατών ε, μας βρίσκει σύμφωνος, είναι καλή ιδέα. Και στη σύγχρηματοδότηση που δεν είναι κρίσιμα σημασία για μας, αλλά μπορεί να είναι για άλλες ομάδες. 90% νομίζω μπορούμε να δεχθούμε. Για να ακολουθήσουμε και την πρόταση της κυρίας Χολμπάια. Σε κάποιες λύσεις λοιπόν μπορούμε να συμπλέψουμε, σε κάποιες άλλες έχουμε απόκληση ακόμα, αλλά ελπίζουμε να σας πείσουμε. Και η δείκτες, όπως είπα, είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικοί. Ευχαριστώ την κυρία Κέλλερ. Εάν θέλει η Επιτροπή, παρακαλώ, να λάβει το λόγο. Για την παρατηρήση της κυρίας Κέλλερ, για τη διαφάνεια. Βεβαίω, η πρόταση της Επιτροπής ε, λέει να καθίσατε να δημοσιοποιείτε η έκθεση στο σύνολό της. Υπάρχουν όμως κάποιες ανησυχίες. Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται σε αυτήν ευαίσθητες πληροφορίες. Θα δούμε. Ίσως αυτό εννοεί το ΕΛΚ. Πάντως για την ε, Επιτροπή πρέπει να είναι δημόσιο. Ε, πρέπει να είναι δημοσιοποιήσιμα τα στοιχεία αυτά, εκτός ίσως από ένα πολύ αυστηρά περιορισμένο ε, αριθμό τους που για συγκεκριμένους λόγους θα μπορούσε να παραμένει απόρριτος ώστε να μην τίθεται σε κινδυνό η ασφάλεια. Αλλά πάντως η βασική αρχή είναι η έκθεση αξιολόγησης να καθίσταται δημόσια. Η αδίποτε παρέκκληση από την αρχή αυτή θα πρέπει να είναι πολύ αυστηρά περιορισμένη. Ο κύριος Φοντάνα έχει το λόγο. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Μου φάνηκε να κατάλαβα ότι θα έχουμε μία νομική γνώμη για να έχουμε σφαιρική εικόνα του πράγματος. Πολλά σημεία χρειάζονται συμφωνία και εγώ πιστεύω ότι το 90% είναι μία σωστή, ένας πολύ σωστός συμβιβασμός. Θα έπρεπε όμως μερικές φορές να φτάνουμε και στο 100% ακούγοντας τώρα τα διάφορα σημεία της ε, Κομισιόν, σίγουρα αυτά θα μας βοηθήσουν να βρούμε μία καλή επαφή με, τον, ε, με τους και εισηγητές. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τη Γραμματεία για τη βοήθειά της αυτές τις τελευταίες μέρες. Ευχαριστώ και εσάς κύριε Φοντάν. Ευχαριστούμε φυσικά τη Γραμματεία. Ευχαριστούμε όλους όσους συμμετέχετε σε αυτή τη συζήτηση που επιβιώσατε αυτές τις ε, πολλές μέρες. Και θέλω τώρα να αναγγείλω τον, ε, την ψηφοφορία 26 και 27 Νοεμβρίου Και αν δεν υπάρχουν διάφορα, Πέντε και 6 Νοεμβρίου επόμενη συνεδρίαση της ΛΥΜΠΕ. Θα τα πούμε την επόμενη φορά.